E- ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να ξεκινήσουμε τώρα τον γύρο ερωτήσεων. Πινκ πόγκα. Ο κύριος Πίτα Λίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε. Ευχαριστώ για την ε, στεναρή δήλωσή σας. Η δήλωση πόθεν έσχες είναι σωστή και μπορώ να διευκρινίσω αγαπητοί φίλοι, κυρία Φαν Μπρέμπτ, την ερώτησή σας. Έχω ένα email από τον Γενικό μας Γραμματέα Κλάους Βέλε και τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή που λένε ότι υπήρξε ένα λάθος στη διοίκηση του Κοινοβουλίου και γι' αυτό φαίνεται τρεις φορές να υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα το οποίο λύθηκε, δεν έχει να κάνει με τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων Επίσης, είχε την καλοσύνη να μην κατηγορήσει τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να μιλήσω για την κλιματική αλλαγή, κύριε υποψήφια επίτροπε. Ε, δείξατε μεγάλη δέσμευση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά ξέρετε ότι ορισμένοι ακόμη και εδώ θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι υπερβολικό, ότι ορισμένοι υπερβάλλουν, ότι δεν υπάρχει ε, καθόλου ε, ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή. Πώς αντιδράτε σε αυτές τις δηλώσεις. Ευχαριστώ για την ερώτηση. νομίζω ότι από το 1988 όταν δημιουργήθηκε το πάνελ IPPC για την κλιματική αλλαγή έχει κάνει θαυμάσια δουλειά. Έχουν κάνει πέντε διαδοχικές ε, αποτιμήσεις ε, κάθε φορά καταδεικνύεται όλο και περισσότερο ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Αυτό είναι σαφές. Πάνω από 2.000 επιστήμονες εργάζονται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών συνεχώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει χρηματοδοτήσει πολλή έρευνα για τους τομείς αυτούς μέσω των προγραμμάτων πλαίσιο. Και τώρα έχουμε το Horizon 2020 που χρηματοδοτεί έρευνα για την κλιματική αλλαγή. Έχουν τεθεί λοιπόν οι αποδείξεις ενώπιόν μας. Οι τρεις ε, τελευταίες δεκαετίες είναι η μία θερμότερη από την άλλη. Από τότε που έχουμε στοιχεία για, την, ε, για, τα, για το κλίμα δεκαετία του 50. Οι ωκεανοί γίνονται πιο ζεστοί, οι πάγοι λιώνουν, τα ακραία φαινόμενα είναι όλο και πιο έντονα. Το βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Δεν μπορούμε λοιπόν να καθυστερήσουμε. Πρέπει να δράσουμε. Πρώτα απ' όλα να τονίσουμε ότι ισχύουν αυτές οι εκθέσεις των επιστημόνων και μετά να τις μετατρέψουμε σε πολιτική δράση. Να αξιοποιήσουμε αυτές τις εκτιμήσεις για να έχουμε φιλόδοξους στόχους στην ε, επικείμενη συνάντηση κορυφής στο Παρίσι. Και πρέπει επίσης να κάνουμε μια τεράστια επικοινωνιακή δουλειά έναντι της κοινή γνώμης. Γιατί αυτοί που αντιδρούν και αρνούνται την ε, κλιματική αλλαγή είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολλές δυνατότητες, ενώ εμείς που ε, στηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει δράση, πολλές φορές ε, είμαστε υπερβολικά επιφυλακτικοί. Θα κάνω λοιπόν πολλές ομιλίες τονίζοντας ότι ε, οφείλεται σε εμά η κλιματική αλλαγή και δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακος, είναι επίσης και το υδρογόνο, διάφορα οξύδια του υδρογόνου και το μεθάνιο. Και θα είμαι πολύ ενεργός προς αυτή την κατεύθυνση. Συγγνώμη, οξύδια του αζότου. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Φαν Μπρέντ. Ευχαριστώ. Κύριε Λίζα, έτσι κι αλλιώς θέλουμε να περιμένουμε την αξιολόγηση της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων. Δεν το χρειάζομαι το μέλη σας. Κύριε Υποψήφια Επίτροπη, για την ε, δήλωση σύγκρουσης εφερόντων θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Πολύ πρόσφατα ανακοινώσατε ότι πουλήσατε τις μετοχή σας στην πετρολίφερα Ντούκαρ και την πετρολίγης Κανάρια. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν να σας κάνω και θέλω απάντηση με ναι ή όχι. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο γιος σας πριν από λίγες μέρες ήταν μέλος του Δικαιωτικού Συμβουλίου και στις δύο αυτές επιχειρήσεις, ότι ο γαμπρός σας σας αντικατέστησε στην Προεδρία και των δύο αυτών εταιριών και είναι αλήθεια ότι η δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη ε, μέτοχη της Πετροφιλέρα είναι εκείνοι που πήραν μέρος αυτών. Μπορείτε επίσης να μας διασφαλίσετε ότι θα τηρήσετε τις υποσχέσεις σας. Εσείς είπατε ότι ποτέ δεν θα ασχοληθώ με θέματα του χαρτοφυλακίου μου εφόσον συγκρούονται αυτά με συμφέροντα που έχουν να κάνουν με την οικογένειά μου. Κλείνει το μικρόφωνο της κυρίας Βαν Απάντηση. Θα σας τα διευκρινίσω όλα. Πρώτα απ' όλα, Με το που έμαθα ότι είμαι υποψήφιος επίτροπος για θέματα ενέργειας, φρόντισα να πουλήσω τις μετοχές μου και παρετήθηκε ο γιος μου. Δεν έχουν μετοχές ούτε θέσεις. Ούτε σε αυτήν την επιχείρηση, ούτε σε καμία άλλη επιχείρηση που να έχει σχέση με αυτήν. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Αλλά ας το δούμε κι αλλιώς. Γιατί δηλώνω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και γιατί γιατί οι δύο αυτές επιχειρήσεις είναι δύο μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 50 εργαζόμενους είναι μικρές. Στα λογιστικά. Δεν κάνουν ούτε εξόριξη πετρελαίου, ούτε πουλούν καύσιμα, ούτε κάνουν επιθεωρήσεις εξορίξεων κλπ. Τίποτα από όλα αυτά. Πρόκειται για δύο μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει λοιπόν σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά προκειμένου να τα σχεδιάσω όλα καλά, πήγα ακόμα πιο μακριά. Πούλησα τις μετοχές μου και ο γιος μου παρετήθηκε. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο γιος μου έχουν θέσει σε επιχειρήσεις αυτές. Ούτε σε καμιά άλλη επιχείρηση που να έχει σχέση με αυτές τις δύο επιχειρήσεις. Άρα δεν υπάρχει κανένα συμφέρον τη οικογένεια μου στι επιχειρήσει αυτέ. E Τώρα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Κύριε Κανιέτα, 40% των στόχων μας για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2020 δεν είναι επαρκές. Και επειδή η σημασία του να έχουμε υποσχέσει ότι θα γίνουν ε, μειώσεις και από όλους μας τους εταίρους ε, στην ε, πορεία προς αυτήν την φάρσα του Παρισιού θεωρείτε ότι θα πρέπει μετά την συνάντηση αυτή θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη, ένα άλλο καθορισμό των στόχων μετά τη συνάντηση στο Παρίσι. Πρώτον, θεωρώ ότι η πρόταση που είναι στο πακέτο για το 2030 είναι ισορροπημένη. 40% μείωση, 25% ανανεώσιμες και 30% ενεργειακή απόδοση. Που ο, Γιούνκερ είπε ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι είναι το ελάχιστο απαραίτητο, το απόλυτο ελάχιστο και θέλει να είναι δεσμευτικό. Είναι λοιπόν ένα συνολικό και ισορροπημένο πακέτο. Θα χρειαστούν λοιπόν πολλέ προσπάθειες από όλους τους τομείς, από όλους τους Ευρωπαίους για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Εάν εμεί φτάσουμε σε αυτή τη συνάντηση κορυφής και όλες οι άλλες οικονομίες του κόσμου, όλοι οι άλλοι μεγάλοι ε, όλες οι άλλες μεγάλες οικονομίες που εκπέμπουν συμφωνήσουν σε πιο φιλόδοξους στόχους Φυσικά δεν θα ήμουν κατά. Φυσικά η Επιτροπή δεν θα έχει αντίρρηση, δεν θα μπλοκάρει πιο φιλόδοξους στόχους. Αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, θα το δούμε. θα δούμε πώς θα συνδυαστεί με το στόχο του 40% για τα διεθνή πιστοποιητικά. Και επίσης ε, πρέπει να δούμε τι ήδη διεθνή πιστοποιητικά και τι ήδη διεθνείς πιστώσεις θα μπορούσαμε να έχουμε στη διεθνή αγορά και τι ποιότητα για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Γιατί δεν ήταν σαφής πάντα η κατάσταση με αυτούς τους καθαρούς μηχανισμούς ανάπτυξης. Ξέρω ότι θα έχω την υποστήριξή σας αν γίνω επίτροπος και θα εξετάσω πολύ προσεκτικά να δούμε τι ποιότητα θα έχουν αυτά τα διεθνή ε, πιστοποιητικά ή διεθνείς πιστώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε. Το χαρτοφυλάκιο, εδώ κάθομαι, για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, ίσω είναι το πιο σημαντικό από ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήμουν υπέρ του να συγχωνευτούν τα δύο αυτά χαρτοφυλάκια. Αλλά εφόσον η Επιτροπή πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και συνδυαστεί η ενέργεια με την κλιματική αλλαγή, ναι, μπορεί μάλιστα να επιτρέψει μεγάλη πρόοδο, αν πάρουμε σοβαρά την πρόκληση αυτή. Οπότε, η ερώτηση σήμερα είναι εξή. Εσεί, κύριε Κανιέτη, είσαστε ο κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβετε αυτό το χαρτοφυλάκιο δεδομένου ότι τα συμφέροντα είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να γίνουν οι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν. Εσεί, λοιπόν με το παρελθόν που έχετε, με τι σχέσει σα με τι πετρελικές εταιρείε, δεν φαίνεται να είσαστε ο σωστό άνθρωπο. Ένα τρόπος υπάρχει για να με πείσετε εμένα και την ομάδα μου ότι είσαστε ο κατάλληλο άνθρωπο. αν μα δείξετε πόσο σοβαρά παίρνετε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πείστε με λοιπόν για το προσωπικό σας αίσθημα για το ότι επήγει να γίνουν οι αλλαγές αυτές για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Απάντηση. Θα προσπαθήσω να σας πείσω. Αλλά πώς να σας πείσω. Κοιτάξτε. Ήμουνα υπουργό περιβάλλοντος στην Ισπανία πριν. Τότε είχα τις μετοχές μου σε αυτές τις δύο μικρές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, πολεμούσα με την ε, Επίτροπο για το Περιβάλλον. Στο πλευρό της. Προκειμένου να προχωρήσουμε με το πακέτο 2030 για πολύ φιλόδοξους στόχους. Ήμουνα και μέρος της ομάδας Green Road στην Ισπανία. Δεν στήριζα το πετρέλαιο, αλλά τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, την, ε, ε, τον φοδιασμό ενέργειας, Έχω ήδη δουλέψει και πολεμήσει για να προστατεύσω τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Δουλεύουμε έτσι καλώ από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να έχουμε ομόφωνες συμφωνίες ουσιαστικά. Πρέπει 200 χώρες περίπου να συμφωνήσουν. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε χρέος στις επόμενε γενιές. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να σκέφτονται βραχυπρόθεσμα, πρέπει να σκέφτονται μακροπρόθεσμα. Η κλιματική αλλαγή απαιτεί μακροχρόνιες, μόνιμες πολιτικές. Είμαι λοιπόν υπέρ αυτών και κατά το παρελθόν. Ποτέ δεν είχα συνδέσει με το πετρέλαιο, είχα ένα 2,5% σε αυτές τις εταιρείε. Όταν όμω είχα δημόσια ευθύνη και δημόσια καθήκοντα, δούλευα υπέρ των ελλακτικών πηγών ενέργειας, υπέρ της ασφάλειας εφοδιασμού. Αυτά κατά το παρελθόν και αυτά θα συνεχίσω να κάνω και στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος Ροντρίγες Ρούμπιο τώρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Κύριε Άρια Κανιέτα, πραγματικά Έρχομαι σε δύσκολη θέση που θα πρέπει και εγώ να μιλήσω για την οικογένειά σας. Αλλά το κάνω γιατί είναι απολύτω απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν έχετε οικογενειακά συμφέροντα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιό σας. Πολύ σπεσμένα ε, πουλήσατε τις μετοχές σας στις πετρελαϊκές εταιρείες Ντούκαρ και, και Αλλά ο κουνιάδος σας έχει άμεση σχέση με τις εταιρείες αυτές. Δεν μας μιλήσατε προηγουμένως ε, για αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνος ε, συνεχίζει να έχει ε, σημαντική θέση στις δύο αυτές πετρελαϊκές εταιρείες. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα φίλο μου που είχε σπουδάσει τοπογράφος πριν την στεγαστική κρίση. Τελικά ασχολήθηκε με τους ηλιακούς θερμοσαρευτές αλλά η κυβέρνησή σα τότε καταπολέμησε τι ανανεώσιμες πηγές ενέργεια ε, και δώσετε έμφαση στις ε, βιομηχανίε εξόριξη. Και ε, ήσασταν κατά της αυτοκατανάλωσης. Ουσιαστικά επιβάλλετε κυρώσει έμεσα με την πολιτική σα Διακόπτει ο Πρόεδρος. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν, σε καμία περίπτωση δεν πώλησα εσπευσμένα τις μετοχές μου. Την Τετάρτη έμαθα από τον πρόεδρο Γιούνκερ ότι θα με προτείνει ε, για τη θέση του Επιτρόπου για το κλίμα και την ενέργεια και την ίδια στιγμή αποφάσισα να πουλήσω τις μετοχές μου για να εξασφαλίσω τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και ανεξαρτησία και να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία, καμία βιασύνη, μόνο διαφάνεια. η ακρόαση αυτή θα κρίνει αν είμαι κατάλληλος και επαρκής για, επί, επίτροπος. Οι επίτροποι είναι απολύτως ανεξάρτητοι από τις εθνικές πολιτικές. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπόλογοι προς τις κυβερνήσεις μας. Εμείς προασπίζουμε το κοινοτικό, το ενωσιακό συμφόρον. Τώρα, αν η Ισπανία υιοθετεί σφαρμένη πολιτική, εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το θέμα. Θέλω να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρωταγωνιστή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλω να τροποποιήσω τις, τα δίκτυα μεταφορών για να μπορέσουν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να βρουν μια διέξοδο εκεί. Και θα σας δώσω και ένα αριθμό αν θέλετε. Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ισπανίας είναι 16,1% το 2013. Ο στόχος είναι 20% για το 2020. Η Ισπανία δηλαδή είναι από τις χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σωστό δρόμο γιατί έχει υψηλό στόχο για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα. Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, η αναζήτηση των καλύτερων πολιτικών. Και επίσης ένα ενιαίο, ομοιόμορφο ευρωπαϊκό σύστημα στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια για να μην δημιουργηθεί στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και να μην τροχοπεδίσουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Και αυτό θα το κάνουμε με τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Eichhout έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, πρώτα απ' όλα. Μπορείτε παρακαλώ να είσαστε σαφέστερος για το γαμπρό σας και τι σχέση έχει με τις διάφορες αυτές επιχειρήσεις. διότι δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Και έπειτα, δεύτερον, κάθε φορά σας παίρνει χρόνο για να αποκαλύπτετε νέα. Όταν, ας πούμε, για την Πετρόλογης ε, Κανάρια το 2011 πήγαν χρήματα, εσείς ήσασταν πρόεδρος της εταιρείας αυτής και μόνο όταν αποκαλύφθηκε το 2014 είπατε ότι δεν το ξέρατε, δεν ξέρατε αυτή τη συμφωνία. Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρατε αυτή τη συμφωνία εφόσον ήσασταν πρόεδρος. Και το ίδιο και με τις μετοχές. Το ακούσαμε ότι μόλις ε, γίνατε υποψήφιος επίτροπος τις ε, πουλήσατε. Γιατί. Μόνο όταν ήσασταν ε, υπεύθυνο για την ενέργεια και το κλίμα. απάντηση. Όσο δεν είχα οριστεί υποψήφιος, δεν είχα κανένα λόγο να τις πουλήσω τις μετοχές αυτές. Είναι μια νόμιμη δραστηριότητα στην Ισπανία. Μόλις έμαθα ότι ήμουν υποψήφιος επίτροπος, ήμουν έτοιμος να τις πουλήσω, ξέροντας ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφέροντος βασικά καθόλου. Αλλά προκειμένου να μην υπάρχει οποιαδήποτε πόνο, πήγα και ακόμα πιο μακριά. Για να μην υπάρχει ακριβώς θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Αποφάσισα, παρόλο που δεν ήμουν υποχρεωμένος, να τις πουλήσω και παρετήθηκα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν συμπληρώνει κανείς τη δήλωση αυτή, οικονομικών συμφερόντων και τον κώδικα διοντολογία σα ρωτάνε ποια είναι τα συμφέροντά σα, τα δικά σα και τη γυναίκα σα. Σα το λέω λοιπόν ότι ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο γιο μου, ούτε εγώ έχουμε κανένα συμφέρον σε καμία επιχείρηση. Είναι σαφέ. Τώρα τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι η στενή οικογένεια. Αυτό ρωτάνε. Και σας απάντησα γι' αυτό. Και το ξέρετε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έδρασα μόλι έμαθα ότι ήμουν υποψήφιο επίτροπο. Όχι νωρίτερα γιατί νωρίτερα δεν μπορούσα. Έτσι και αλλιώ χρειάζονται τρει με πέντε μέρε στην Ισπανία για να πουλήσει μετοχέ. Δεν μπορεί να το κάνει αμέσω, γιατί πρόκειται για μια ιδιωτική περιορισμένη επιχείρηση. Με απόλυτη διαφάνεια λοιπόν προχώρησα και πήγα και ακόμα πιο μακριά από αυτό το οποίο μου ζητάτε. Και νομίζω ότι είμαι σαφή όταν λέω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι η οικογένειά μου, η γυναίκα μου και ο γιος μου δεν εμπλέκονται στις επιχειρήσεις αυτές, ούτε και σε καμία άλλη επιχείρηση που έχει να κάνει με πετρέλαια. Ευχαριστούμε. Συνάδελφος Πεντιτσίνη τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Καλησπέρα κύριε Κανιέτε. Μέχρι στιγμή μιλήσαμε για την οικογένειά σα. Εγώ θα σα μιλήσω για τη δική μου οικογένεια. Γιατί και εγώ και η οικογένειά μου και όλο ο λαός, όλοι οι συμπολίτε μου ζούμε σε μια περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί που χρησιμοποιείται υδρορογμάτωση για την εξόριση πετρελαίου εδώ και 20 περίπου χρόνια. Έχω λοιπόν εύλογους λόγους για να σας πω ότι στην πατρίδα μου έχουμε τεράστιο ποσοστό ανεργίας και νέων και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να καταστρέφουμε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να τις διαθέσουμε σε εξοριστικές βιομηχανίες. Για να μην μιλήσω για τα απόβλητα που δημιουργούν αυτές. Και επίσης έχουμε αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου που οφείλονται σε βαρέα μέταλλα ή σε εισπνοή τοξικών αερίων. Τι λοιπόν θα κάνετε για τη δημόσια υγεία, γιατί η ενθάρρυνση τέτοιων βιομηχανιών αποβαίνει μοιραία για την υγεία των πολιτών. Όπως ξέρετε, κύριε Βουλευτά, η συνθήκη εκχωρεί το αποκλειστικό δικαίωμα στα κράτη-μέλη να εκμεταλλεύονται και να διαχειρίζονται όπως επιθυμούν τον ορυκτό τους πλούτο και τις πηγές ενεργειάς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλε συστάσεις χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα προβλέποντας ότι σε περίπτωση που λυθεί σχετική απόφαση, η εξόριξη θα πρέπει να γίνεται με βάση κάποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν σύσταση έχει υποβάλει, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως έχει τεθεί σε ισχύ ένα δίκτυο, ένα επιστημονικό δίκτυο, που θα αναλύσει όλες τις εμπειρίες εξόρυξης και σχιστολιθικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη για να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και οι συνέπειες για το περιβάλλον αυτής της μορφής εξόρυξης. Επίσης θα μπορούσα να προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την εξόριξη σχιστολιθικού αερίου με βάση συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον αρμόδιο επίτροπο περιβάλλοντος. Σας διαβεβαιώ ότι θα συγκεντρώσουμε και θα αναλύσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, τις συνέπειες τους στα οικοσυστήματα, στους υδροφόρους ορίζοντες, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες και με βάση αυτή την ανάλυση θα κρίνουμε αν είναι σκόπιμο να θεσπίσουμε δεσμευτικές διατάξεις για να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό. Το θέμα δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί επαναλαμβάνω υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών για το θέμα αυτό αλλά έχουμε και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαφυλάξει το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τα φυσικά ενδιατήματα, τους υδροφόρους ορίζοντες και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Πιλάρ Δελκαστήλιο κύριε υποψήφια επίτροπε κύριε Αρία Κανιέτε. Ευχαριστώ για την σαφήνεια και την ε, αφοσίωση που ακούσαμε στην ομιλία σας για την κλιματική αλλαγή και για την ενέργεια. Σίγουρα θα επιμείνουν διάφοροι σε κάποια οικογενειακά ζητήματα σε όλη τη διάρκεια της συζήτηση. Γιατί εφόσον απεδείχθη ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, γιατί και ορισμένα πράξατε εσείς αλλά και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τα έλεγξε οπότε να περάσουμε στην ουσία. Εγώ θέλω να μιλήσω για θέματα ενεργειακής ανεξαρτησίας. Φυσικά η έλλειψή της οφείλεται σε έλλειψη και υποδομών που δημιουργεί αυτούς τους δίλακους και Επίσης μπορεί να βοηθήσει ανάπτυξη των ευφυών δικτύων. Έχουμε πολλά ε, προγράμματα που έχουν υποβληθεί και δεν έχουμε επαρκές πιστώσεις. Τι θα αξιοποιήσετε εσείς για να πιέσουμε να υπάρξει εξυγχρονισμός των δικτύων και να υπάρξει η αναγκαία διασύνδεση των δικτύων που είναι απαραίτητη. Προφανώς. Για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια χρειάζονται διασυνδέσεις στη Βαλτική, στην Ιβυρική Χερσόνησο, στην Ανατολική Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο, ενοποιημένο και ευφυές δίκτυο που να το, μας επιτρέπει να αξιοποιούμε πλήρως ε, αυτές τις διασυνδέσεις. Η ελάχιστη δέσμευση που συμφωνήθηκε στην Βαρκελόνη το 2000 υπήρχε ένας ενδεικτικός στόχος 10% ε, ελάχιστο διασυνδέσεων. Ο στόχος αυτός ε, βεβαίως έχει εκπληρωθεί και με τα προγράμματα ενωσιακού συμφέροντος ε, θα προχωρήσουν για το φυσικό αέριο και την ενέργεια. Δυστυχώς υπάρχει μία εξαίρεση που μας ε, λυπεί ιδιαίτερα, είναι η Βυρική Χερσόνησος που είναι σαν νησί. Και πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και σε αυτό. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή θέλει να ξεκινήσει διάλογος με τις ρυθμιστικές αρχές στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία για να ξεπεράσουμε αυτό το μπλοκάρισμα και υπάρχει ένα πρόγραμμα διασύνδεσης μέσω των Πυρηναίων που ήδη έχει ξεκινήσει ούτως ώστε να περάσουμε από τα 400 στα 800 ΜΒ αλλά ορισμένα άλλα είναι πολύ αργά. Για παράδειγμα να διασυνδεθεί η Ακουιτανία με τον Βυσκαϊκό κόλπο μέσω των Πυρηναίων. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια από την Επιτροπή γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα χρηματοδότηση. Πρέπει επίσης επειδή ε, οι δυνατότητες του διασυνδέοντας στην Ευρώπη δεν είναι αρκετές να δούμε πού αλλού μπορούμε να βρούμε την αναγκαία χρηματοδότηση, για παράδειγμα από τα 300 δις του πακέτου Juncker, για να έχουμε συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρότε. Τις τελευταίες εβδομάδες, κύριε Κανιέτε, η σχέσεις σας ε, και οι οικογενειακοί σας σχέσεις με την ενεργειακή βιομηχανία συζητήθηκαν πολύ και χθες ε, προσαρμόσατε και πάλι τη δήλωσή σας. Καγιοργά παρά ποτέ. Και για το backloading επίσης καθυστερήσατε, αλλά πολύ αργά και αυτό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εκπομπών, το σύστημα ε, εμπορίας εκπομπών. Θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα σταθεροποίησης της αγοράς ή θεωρείτε ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μετά το 2020 όταν ίσως να είναι πολύ αργά για αυτό το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών. Παρακαλώ, ε, είπατε ήδη ορισμένα για την οικογένειά σας. Παρακαλώ, οι στενείς συγγενείς να μας πείτε πώς συνδέονται με αυτές τις επιχειρήσεις. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Γι' αυτό καλύτερα να απαντήσω στα αγγλικά. Δεν επαρκούν τα γερμανικά μου. Πρώτον, θεωρώ ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είναι θαυμάσιο μέσο. Έχουμε ένα σύστημα τιμών για, το, για τα αέρια, άνθρακος, αλλά παρά τα προβλήματά το σύστημα αυτό λειτουργεί. Είναι επαρκές για να μας οδηγήσει σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων άνθρακο. Θέλω λοιπόν αυτό το σύστημα ETS να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αλλά επίση, με ρωτήσατε για το αποθεματικό για τη σταθεροποίηση τη αγορά. Νομίζω πω είναι ευφυές ε, όργανο, ευφυής μηχανισμό. Ε, αποφεύγει αυτά τα πολιτικά παιχνίδια με την τιμολόγηση της ενέργειας. Αν είναι υπερβολικά τα ποσά πάνω στο αποθεματικό, αν είναι ανεπαρκή, παίρνεις από το αποθεματικό και μας επιτρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε. Με ρωτήσατε αν θα πρέπει να προχωρήσουμε ή όχι. Φοβάμαι. Θεωρώ ότι το backloading ήταν ε, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο μια φορά και αυτά που έχουμε αφαιρέσει από την αγορά θα επανέλθουν. Άρα μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές. Και αυτό θα ήταν ε, κακή εξέλιξη. Αν λοιπόν με υποστηρίξετε παρκώς εσείς εδώ, θα επιχειρήσω να πείσω το Συμβούλιο, ούτω ώστε το αποθυματικό για τη σταθεροποίηση της αγοράς να αρχίσει να εφαρμόζεται νωρίτερα. Γιατί αυτό θα αποτρέψει τις ε, στρεβλώσεις της αγοράς και ακόμη και τις διαταράξεις στην αγορά που μπορεί να προκαλέσει η επάνωδος του backloading. Αρκεί να έχουμε την πλήρη υποστήριξή σας για το μέτρο αυτό, γιατί όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι περίπλοκα. Χρειάζομαι λοιπόν την εκ των προτέρων στήριξή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιατσκέβιτς. Ευχαριστώ. Κύριε Κανιέτε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας υποβάλλετε τις ε, πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να, να λάβετε για να ενισχύσετε την ε, ενεργειακή μας ανεξαρτησία ε, και από προμηθευτές, ε, διαδρόμους και διάφορα είδη και πηγές ενέργειας. Ποιες είναι οι προτάσεις που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία. Επίσης, πώς θα στηρίξουμε τις τοπικές αρχές για να αξιοποιήσουν τις πηγές ενέργειάς τους. Τι συνέπεια θα έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην επαναβιομηχάνηση η μεταρρύθμιση που θα προταθεί για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ποιοι βιομηχανικοί τομείς θα υποστηριχθούν από το... και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στους... από το σύστημα εμπορίας εκπομπών όπως θα μεταρρυθμιστεί και ποιοι θα πληγούν από τις αλλαγές αυτές στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ευχαριστώ. First of all, uh... Καταρχάς, πιστεύω ότι για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές ανεφοδιασμού μας. Δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε από ένα και μόνο προμηθευτή για πετρέλαιο και ε, φυσικό αέριο. Και επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε τις διασυνδέσεις μας ανά την Ευρώπη. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τον νότιο διάδρομο. Είναι σαφές ότι το South Stream δεν θα προχωρήσει αν προηγουμένως δεν ε, εφαρμόσουμε το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου. Αλλιώς θα μείνουμε εξαρτημένοι σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και φυσικά να αναπτύξουμε και κάποια προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, θα πρέπει να βρούμε κονδύλια και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Το 20% των διαρθρωτικών ταμείων αφιερώνεται στην καταπολέμηση των, ε, κλιματικών αλλαγών και την ε, διόρθωση προβλημάτων στον ενεργειακό τομέα. Θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια. Επίσης, με ρωτήσατε πώς θα λειτουργήσει το μεταρρυθμισμένο σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS, και πώς θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων της βιομηχανίας θα, πρέπει, θα έχουμε και το σύστημα των ε, δωρεάν αδειών για κάποια κρατημέλη. Των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών. Μερικά κράτη ήδη εφάρμοσαν αυτό το σύστημα και μάλιστα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να δούμε τι αλλαγές θα επιφέρουμε ώστε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ή και να τη βελτιώσουμε. Επίσης, θα πρέπει να ε, στηρίξουμε και τις χώρες που θέλουν να κρατήσουν κάποια ενεργειακά εργοστάσια, είτε ε, εφαρμόζοντας το παλιό σύστημα, είτε προβλέποντας συγκεκριμένες αλλαγές στο νέο σύστημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με δύο μεγάλες προκλήσεις σήμερα. Πρέπει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και πρέπει να βελτιώσει και την ενεργειακή μας ασφάλεια μέσω του ενεργειακού εφοδιασμού με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και μειώνοντας την εξάρτησή μας από εισαγόμενα καύσιμα δεδομένης της δυνατότητας που υπάρχει για μεγαλύτερη παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενεργειών, αιωλική κλπ. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτές οι δυνατότητες που υπάρχουν για καθαρή, βιώσιμη ενέργεια θα ληφθούν πλήρως υπόψη και θα χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς εσείς προσωπικά θα διασφαλίσετε μια πραγματική ενιαία ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη που είναι και το κλειδί για να λυθούν αυτές οι δύο μεγάλες προκλήσεις που έχει η Ευρώπη μπροστά της σήμερα. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα για να αναπτύξουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Το μεγαλύτερο είναι ότι δεν έχουμε ακόμα μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί καλά. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην εσωτερική αγορά. Δεν υπάρχουν δίκτυα, για παράδειγμα, για να παίρνουμε την ε, ενέργεια κλπ. Συνεπώς, πρέπει να επενδύσουμε και προσπαθώ να αναπτύξω νέα νομοθεσία για μια ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Όταν γίνει αυτό θα έχουμε επαρκή δίκτυα. Θα έχουμε φορείς οι οποίοι συντονισμένα θα, θα δρουν και θα μπορέσουμε έτσι να αναπτύξουμε περισσότερο τις δυνατότητές μας. Βέβαια και σε περιφερειακό επίπεδο στη Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα, πρέπει να στηρίξουμε προγράμματα όπως είναι η πρωτοβουλία για τα offshore δίκτυα και άλλα αντίστοιχα προγράμματα. Σε περιφερειακό επίπεδο προς το παρόν μέχρι να έχουμε ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά συστήματα. Άρα χρειάζεται η περιφερειακή ολοκλήρωση, διασυνοριακή συνεργασία και σιγά σιγά να προχωρήσουμε προς την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Πάντως το πρόβλημα με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας θα παραμείνει όσο δεν έχουμε προχωρήσει με τα δίκτυα. Άρα χρειαζόμαστε φύη δίκτυα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Συγχρόνως πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λόμπες Μπερμέχο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Κανιέτε, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας είμαι γυναίκα, πολύ θα ήθελα να κάνουμε αυτό το διάλογο μαζί, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Πάντως, η κυβέρνησή σας κατάργησε τις εναλλακτικέ ενέργειες στην ε, Ισπανία. Είπατε υπέρ του φράκινγκ, της υδρορογμάτωσης, υπέρ του λιγοπολίου του ηλεκτρισμού, αδιαφορώντας για τα εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλετε εσείς για την Ευρώπη. Πώς έρχεστε εδώ σήμερα και μας λέτε το αντίθετο από αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Έπειτα εσείς δεν έχετε καμία νομιμότητα για το χαρτοφυλάκιο αυτό, γιατί υπάρχουν τα συμφέροντά σας. Κάθε μέρα αλλάζανε τα πράγματα. Χτες μάθαμε για την αναμειξή σας στην ε, εκλογική επιτροπή του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος. Δεν μπορούσατε να μας το είχατε πει νωρίτερα. Οι πετρελαϊκές εταιρείε, τα... οι δημόσιες συμβάσεις που έπαιρναν επιχειρήσεις αυτές. Πώς, με ποιο τρόπο. Όλα αυτά όμως περνάνε από μια ε, επιχείρηση στην Ολλανδία. Διακόπτει το μικρόφωνο ο πρόεδρος. Απάντηση. Δεν κατάλαβα ποια ακριβώ είναι η ερώτησή σας. Θα προσπαθήσω όμω παρόλα αυτά να σας απαντήσω. Το είπα και νωρίτερα εδώ. Αν αναλάβω τελικά το χαρτοφυλάκιο, εγώ δεν θα υποστηρίξω καμία εθνική πολιτική, αλλά ευρωπαϊκές πολιτικές υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ανέργειας και διάρθρωσης των αναλλακτικών πηγών ανέργειας να υπάρχει επίσης όρις δράση στην Ευρώπη. Αυτό που έρχομαι εγώ να κάνω στην Ευρώπη είναι να ρυθμίσω την εσωτερική αγορά ώστε να υπάρξουν συστήματα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αποφύγουμε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κάποιες χώρες όπως η Ισπανία, όχι με την κυβέρνηση όπου εγώ συμμετείχα, αλλά με προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες δώσαν υπερβολικές επιδοτήσεις και έκαναν το παιχνίδι να μην μπορεί να παιχτεί τελικά και καταλήξαμε σε τεράστιο έλλειμμα. Γι' αυτό λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που θα κάνουμε είναι να καθορίσουμε κανόνες για να υπάρχει ένα σύστημα στήριξης που να βασίζεται στην αγορά χωρίς να βαραίνει σε επιδοτήσεις από τις χώρες μέλη και να είναι ενιαίος ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό αποτελεί εγγύηση για τον ανταγωνισμό όπως επίσης και με την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων. Σε αυτά θα αφιερωθώ ως Επίτροπος. Να δώσω πρόθεση σε μια φιλόδοξη πολιτική ενεργειακού εφοδιασμού, αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής. Θα στηρίξω μια πολιτική υπέρ των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, υπέρ της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, ώστε η Ευρώπη να γίνει ανεξάρτητη, κάτι το οποίο τόσο πολύ χρειάζεται σήμερα από το φυσικό αέριο και να αποφύγει την απομόνωση που πλήττει κάποιες χώρες. Ευρωπαϊκές πολιτικές λοιπόν θα προσπαθήσω να βρω ό,τι καλύτερο ώστε να αποφεληθούν όλες οι χώρες μέλη, ακόμα και εκείνες που παλιότερα είχαν προβλήματα επειδή υιοθέτησαν λαθασμένες πολιτικές. Ευχαριστώ. Η κυρία Βιβασί. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Κανιέτερ μία από τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η διαφάνεια. Και όταν εξετάσω τις σταδιοδρομία σας ως υπουργό Περιβάλλοντος, δώσατε άδειες εξόριξης στην εταιρεία Rapsol εκ, λίγο έξω από τις ακτές των Καναρίων. Πρώτον, πήρατε, 12, ε, πήρατε δεκάδες αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα από δημόσιες αρχές για να δούμε πώς δόθηκαν αυτές οι άδειες και τις απορρίψατε όλες. Δεύτερο λάθος γίνονται εξορίξεις στη Μεσόγειο, γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, ενώ όλες οι βιομηχανίες, όλοι οι κλάδοι και οι δημόσιες αρχές ήταν κατά οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια. Στα πλαίσια της αναθεώρησης των κανόνων για την αναθεώρηση της ασφάλειας των ε, πλατφορμών εξόριξης, τι ε, εμπιστοσύνη μπορούμε να σας έχουμε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας κυρία μου. Θα σας πω το εξής. Δεν ήμουν ο υπουργό της βιομηχανίας της χώρας μου. Δεν πήρα την απόφαση να δοθεί έγκριση για την εξερεύνηση για πετρέλαιο, γιατί αυτές τις δίνει το Υπουργείο Βιομηχανίας. Το μόνο που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η Ισπανία είναι κράτος δικαίου. Η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται από εμπειρογνώμονες, όχι από πολιτικού. Έχουμε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες που κάνουν αυτές τις ε, μελέτες επιπτώσεων. Εάν είναι θετικές οι μελέτες, τότε χορηγούμε τις άδειε. Αν αρνητικές, τις απορρίπτουμε. Εγώ αρνήθηκα την δημιουργία του μεγαλύτερου διελιστηρίου στην Ισπανία γιατί η μελέτη επιπτώσεων ήταν αρνητική αλλά ποτέ δεν επιχείρησα να επηρεάσω μια τέτοια, ε, μια τέτοια εκτίμηση άφησα τους αρμόδιους υπαλλήλους να πάρουν τις αποφάσεις, διότι αυτοί με βάση επιστημονικά κριτήρια πρέπει να αποφασίζουν. Ή αν οι αποφάσεις για περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται με πολιτικά κριτήρια, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η οδηγία για την ε, εξερεύνηση πέραν των ακτών που ε, πρόσφατα τροποποιήθηκε. Έχουμε ένα σωστό μέσο που διασφαλίζει την ασφάλεια αν υπάρξουν ατυχήματα, έχει όλους τους προληπτικούς μηχανισμούς και συστήματα και θα δω πώς θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα ε, κάνουμε ακόμη πιο αυστηρή την πρόληψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήμουν υπουργό Περιβάλλοντος, άφησα τους εμπειρογνώμονές μου να εκφραστούν και ακολούθησα πάντα τις απόψεις τους. Δεν πήρα καμία πολιτική απόφαση για να στηρίξω ένα φίλο κτλ. Βασίστηκα στην καλύτερη επιστημονική αρρωγή που μπορούσα να έχω και ε, εμπιστεύομαι τους εμπειρογνώμονες, όπως τους εμπιστεύομαι και στα Ηνωμένα Έθνη. Κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος, έληξε ο χρόνος σας. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Χέλμερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, υποψήφια Επίτροπε. Είμαι ο εκπρόσωπος για την ενέργεια της μεγαλύτερης βρετανικής αντιπροσωπείας στο Κοινοβούλιο, εθνικής αντιπροσωπείας. Ξέρουμε ότι δεν έχει υπάρξει 18 χρόνια καμία θέρμανση του πλανήτη, καμία αυτό τον αιώνα. Ξέρουμε επίσης ότι η τρομερή υπερβολική αφοσίωση στις ανανεώσιμες έχει δημιουργήσει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Και το ξέρουμε αυτό γιατί ο Επίτροπος Άιτιγκερ είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πια να πληρώσει μια μονομερή ενεργειακή πολιτική και ο προηγούμενος επίτροπος Τατζάνη είπε ότι οι τιμές ενέργειας δημιουργούν μακελιό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θα κάνετε κάτι για να λύσετε το πρόβλημα. Έχετε κανένα ε, σχέδιο για να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητα. Θα διασώσετε τις οικονομίες μας από αυτήν την συμφορά για την ανταγωνιστικότητά μας που δημιουργήθηκε από τη μονομανία μα με τα πράσινα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω όσον αφορά την θέρμανση. Δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα στατιστικών. Κάθε τρεις ε, δεκαετίες αυξάνεται η θερμοκρασία. Είναι σαφές στοιχείο αυτό. Αυξάνεται η, η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,3 και αν υπερβεί τους δύο βαθμούς ε, αύξηση θα έχουμε καταστροφικές συνέπειες. Πρέπει λοιπόν με βάση αυτήν την θεώρηση να δράσουμε. Βεβαίως έχουμε πρόβλημα με την ε, τιμή της ενέργειας, με τις τιμές της ενέργειας, γιατί δεν έχουμε επαρκής, ε, επαρκή αποθέματα φυσικού αερίου, εξαρτώμεθα από άλλους για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην τιμή της ενέργειας. Οπότε έχουμε πρόβλημα σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αναπτύξουμε τις δικές μας πηγές ενέργειας. Γι' αυτό στηρίζουμε τις ανανεώσιμές μας, υποστηρίζουμε την ενεργειακή απόδοση και πρέπει επίσης να έχουμε περισσότερη διαφοροποίηση πηγών και να αυξήσουμε και τη δυνατότητα μεταποίησης ενέργειας. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε ως Ευρωπαίοι για να έχουμε περισσότερη αγοραστική δύναμη. Διότι αυτή τη στιγμή κάθε εταιρεία συνάπτει τις δικές της συμβάσεις. Ο σύνολο θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερες τιμές. Αν μπορούσαμε να έχουμε μια δυνατότητα από κοινού διαπραγμάτευσης για την αγορά ενέργειας. Θα κάνω ό,τι μπορώ να πείσω τους εμπλεκόμενους να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Συνολικά, τι πρέπει να κάνουμε. Να πούμε ότι δεσμευόμεθα να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, να το πούμε στο Παρίσι και να απαιτήσουμε όλες οι χώρες να αναλάβουν τις ίδιες ευθύνες για να έχουμε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόντιν. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επιτρόπε. Άκουσα κι εγώ και είμαι επιφυλακτική ως προς τη πιθανή σύγκρουση φερόντων που σας αφορά γιατί δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, όπως λέμε στη Γαλλία. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις, ε, ε, στις υπεράκτηρες ε, ανεμογεννήτριες, παρόλο που τα περιβαλλοντικά τους αποτελέσματα είναι αμφισβητήσιμα. Και από οικονομική άποψη δεν αναπτύσσονται όπως περιμέναμε. Σήμερα η αποτυχία ενός σχεδίου στη Βόρεια Θάλασσα δείχνει ότι η μεγάλη κλίμακος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες είναι ανέφικτη. Ερωτώ λοιπόν, θα ζητήσετε ανάλυση οικολογικών και οικονομικών επιπτώσεων των ανεμογεννητριών, ιδιαίτερα των υπεράκτιων ανεμογεννητριών και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας θα ήθελα να πω ότι είναι καλό να συγκεντρώνουμε στοιχεία από όλα μας τα προγράμματα και να τα αναλύουμε για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Αλλά έχουμε πρόβλημα έλλειψης ενέργειας, ε, λοιπόν διασυνδέσεων και μεγάλα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα στη Βόρεια Θάλασσα, ε, δίκτυα υπεράκτια, προσπαθούν να συνδυάσουν διάφορες προσπάθειες και να αναμίξουν και τις περιφερειακές αρχές. Όχι μόνο για να έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το θέμα αυτό αφορά και το backup, το μηχανισμό backup, αλλά και το φυσικό αέριο. Και θέλουμε να λύσουμε το μείζον ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις όλων των ευρωπαϊκών σχεδίων και προγραμμάτων. Και αναλαμβάνω τη δέσμευση να ζητήσω μελέτες επιπτώσεων για όλα τα προγράμματα και τα σχέδια που θα προτείνω. Επιπτώσεων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών. Σας υπόσχομαι ότι για όλα τα σχέδια που θα υποβάλω θα ζητήσω προηγούμενη τέτοια μελέτη επιπτώσεων. Και επίσης ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Χρειαζόμαστε τέτοια ευρία διαβούλευση, ευρύ διάλογο και φυσικά μελέτες επιπτώσεων για να δούμε πώς επηρεάζουν συγκεκριμένα σχέδια την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ πάντως ότι όλες αυτές οι πτυχές θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρινς. Ευχαριστώ, κύριε Προτινόμενε Επίτροπε. Το χαρτοφυλάκιο κλιματικές δράσεις και ενέργεια ε, εμπεριέχει έναν κίνδυνο γενή και ένα δίλημα. Έχουμε τη συλλογική ανάγκη μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και τη επιβράδυση των κλιματικών αλλαγών. Απ' την άλλη, έχουμε το συμφέρον των καταναλωτών και τη βιομηχανία για χαμηλό ενεργειακό κόστο, αύξηση τη ανταγωνιστικότητα και αύξηση των θέσεων απασχόληση. Ερωτώ λοιπόν, Ποιος κατά τη γνώμη σας θα είναι ο ρόλος σας για την, να βρείτε αυτή την ισορροπία δεδομένη στις ανάγκες και της ενεργειακής ασφάλειας, δηλαδή της μείωσης της ενεργειακής μας εξάρτησης από εισαγόμενο αέριο και μάλιστα από τη Ρωσία. Πιστεύω ότι ίσως αυτό θα είναι το πιο δύσκολο δίλημα, γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ενεργειακό ενεφοδιασμό για όλους τους Ευρωπαίους, αλλά σε λογικές τιμές, σε προσιτές τιμές. Και εδώ δεν αρκεί μία και μόνο δράση, αλλά πολλές δράσεις σε πολλά επίπεδα. Θέλουμε ενεργειακή απόδοση, γιατί με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έχουμε και οικονομίες, αλλά και πιο εύκολα θα εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια. Λοιπόν, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, έχουμε την σχετική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Βέβαια, οι διατάξεις θα ισχύσουν μετά από το 2020. Τι θα γίνει με, την, με το οικολογικό design και την, ε, την επισήμανση, την, ενέργεια την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Επίσης, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλουμε να έχουμε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, φθηνότερες τιμές. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακόμη δεν έχουν αξιοποιήσει όλες τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα είναι σημαντικό, το CCS. Και φυσικά εξασφάλιση διασυνδέσεων. Και ο νότιος διάδρομος αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα. Θα πρέπει να έχουμε διασύνδεση και της Βαλτικής βέβαια και αυτή είναι απαραίτητη και θα δούμε τι θα γίνει με τον συγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων. Δαπανηρό εγχείρημα, αλλά το χρειαζόμαστε. Είναι απαράδεκτο τρεις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι συγχρονισμένες με το ευρωπαϊκό σύστημα. Όλες αυτές οι δράσεις θα γίνουν παράλληλα. Αλλά θα πρέπει και οι ανταγωνιστές μας, οι εταίροι μας να εστερνιστούν αυτές τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές για να μην έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού. δεν είναι εύκολο πάντως να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ των χαμηλών ενεργειακών τιμών και τον, ε, του στόχου των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Μάρτιν Έντουαρτ. Κύριε Κανιέτα, ήσασταν υπουργό όταν η Ισπανική κυβέρνηση 30 Οκτωβρίου 2013 νομιμοποίησε την υδρορογμάτωση και ξεκίνησε τις ε, εξερευνήσεις για σχιστολιθικό αέριο. Και επίσης εγκρίνατε την πρώτη μεγάλη παράδοση καναδικών σχιστολιθικών άμμων στην Ισπανία. Θεωρείτε λοιπόν ότι η υδρορογμάτωση είναι τόσο ακίνδυνη και είναι δυνατόν να την επιβάλλουμε στον πληθυσμό μας. Ενώ παντού στην Ευρώπη γίνονται διαδηλώσεις κατά της δρορογμάτωσης, ε, γίνεται συλλογή υπογραφών. Και εδώ δεν επιτρέπεται από την κυβέρνηση η δρορογμάτωση. Πώς καταλήξατε σε άλλη άποψη στην Ισπανία και η διάσκεψη του Παρισιού που επίκειται. Μπορείτε να μας πείτε τι ύψος αερίων θερμοκηπίου που θα προκύψουν από την ε, ε, χρήση αυτών των μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η απόφαση να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες υδρορογμάτωσης και σχιστολιθικό αέριο είναι ευθύνη των ε, εθνικών κυβερνήσεων με βάση τις ε, συνθήκες. Άλλες κυβερνήσεις μπορούν να το επιτρέψουν και άλλες μπορούν να το απαγορεύσουν. Η Επιτροπή έκανε μία σύσταση. Εάν επιχειρήσουν να κάνουν υδρορογμάτωση, τι κατευντήρες γραμμές πρέπει να σεβαστούν όσοι ζητούν άδειε. Δεν ήμουν εγώ υπουργό που ενέκρινε την υδρορογμάτωση. Ω υπουργό, πριν τη σύσταση τη Κομισιόν, ω υπουργό λοιπόν αποφάσισα ότι η υδρορογμάτωση θα υπόκειται στις πιο αυστηρές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή ήταν η απόφασή μου, ότι η υδρορογμάτωση θα πρέπει να είναι αντικείμενο περιβαλλοντικών μελέτης επιπτώσεων με τα πιο αυστηρά, τα πιο σκληρά κριτήρια. Τώρα η Κομισιόν έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο για να δει τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Και με βάση ό,τι θα μάθουμε ουσιώδη επιστημονική, πρακτική επιστημονική γνώση, τότε αν αναγκαίο θα προτείνω την κατάλληλη νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Στη συνάντηση κορυφής στο Παρίσι, τι θα κάνουμε. Θέλουμε μια δεσμευτική συμφωνία όλων των χωρών που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις. Να δούμε σε ποιο κοινό έδαφος θα μπορούσαμε να καταλήξουμε. Εμείς είμαστε πρωτοπορία γιατί θα εγκρίνουμε τον Οκτώβριο ένα πολύ ουσιώδες πακέτο και το 40% είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος που προτείνουμε. Ευχαριστώ κύριε Βυσνιεύσκα. Σας ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ, ε, ε, εκπέμπει λιγότερο από το 10% των παγκόσμιων ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μάλιστα θα μειώσουμε στο 4% το 2030. Τι πρόκειται να κάνετε στα πλαίσια του μελλοντικού ενεργειακού κλιματικού πακέτου μέχρι το 2030 προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιβίωση των ενεργειοβόρων βιομηχανιών που είναι όμως απαραίτητες για την ε, επιβίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η γεωπολιτική κατάσταση και συγκεκριμένες ε, πρώτες ύλες. Μόνο έτσι ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους στόχους αναλογικά με τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, πώς ε, θα, θα πείσουμε τους εταίρους μας όπως η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε που είναι οι, από τις χώρες που εκπέμπουν περισσότερες, περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου να μειώσουν αυτές τις εκπομπές. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε για να συμμορφωθούμε με τους στόχους μας ε, για την ενέργεια και το περιβάλλον είναι να εφαρμόσουμε τους στόχους ε, για το 2020. Γιατί έχουμε νομοθεσία, θα πρέπει να την εφαρμόσουμε με τους στόχους που έχουμε θεσπίσει. Γιατί πολλά, πολύ νερό θα περάσει από το βλάκι μέχρι το 2020. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους στόχους αυτούς στον διάμεσο διάστημα. Θα έχουμε την οδηγία για την ενίσχυση του ETS, του συστήματος Εμβορίας εκπομπών και επίσης ε, τι θα κάνουμε και οι εταίροι μας που εκπέμπουν ε, ε, αέρια του θερμοκηπίου να αναλάβουν και αυτοί και να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο θα έχουμε διπλωματικές επαφές με τους εταίρους μας. Θα έχουμε συνεχείς τακτικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο σημαντικό οικονομικό φόρουμ που είναι σημαντικό για τις ανεπτυγμένες χώρες που εκπέμπουν και πολλές εκπομπές. Θα θέσουμε το θέμα και στο G7 και στο G20 για να ετοιμάσουμε τις δεσμεύσεις και φυσικά και οι διμερείς επαφές θα έχουμε με την Ινδία, την Κίνα που είναι σημαντικοί παγκόσμιοι παράγοντες αλλά και με τις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί και αυτές θα πρέπει να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για το κλίμα των Παρισίων. Οπότε θα έχω επαφές και με λατινοαμερικανικές χώρες, με την ομάδα ΦΕΙΛΑΚ ώστε να υιοθετηθούν στο Παρίσι δεσμευτικοί στόχοι. Είναι σημαντικό να αναλάβουν όλες οι χώρες του κόσμου δεσμεύσεις για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστούμε, η κυρία Μπέρνερ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, είμαι γυναίκα, αλλά θα σας κάνω μια περίπλοκη ερώτηση. Το να πετύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία για την μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι ζωτική σημασία για να αποφύγουμε την κλιματική αλλαγή. Οι αιτίε όμως είναι πολύ ευρειε και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, έχει να κάνει με την ε, αποψήλωση, έχει να κάνει με άλλα θέματα όπως είναι μετανάστευση κτλ. Τι λοιπόν στρατηγική θα ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις αυτές και μην ξεχνάτε ότι όλε οι χώρε του κόσμου περιμένουν την Ευρώπη να έχει τον ηγητικό ρόλο. Λέτε ότι θέλετε η Ευρώπη να αποτελέσει, να αποκτήσει μάλλον ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση των κλιματικών αραγών. Ε, δεσμεύεστε και για δεσμευτικές ε, προτάσεις και μετά το 2020, ώστε όλοι να τηρήσουν τους κανόνες και να αποφεύγεται η αποψήλωση στις ε, υποανάπτυξη χώρες, για παράδειγμα. Και η λοτομία. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα θα αναλάβω δράση σε όλους τους τομείς. Γιατί θα συνεργαστούμε και στο Λούλου και σε όλους εκείνους τους τομείς, γεωργία, μεταφορές, τα πάντα. Και αν θέλουμε μια φιλόδοξη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, πρέπει να βοηθήσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προκειμένου να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Μια από τις, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στο Παρίσι θα είναι το οικονομικό πακέτο. Πώς θα πετύχουμε δηλαδή συμβασμούς με τις χώρες αυτές. Διότι εμείς έχουμε δεσμευτεί. 100 εκατομμύρια δολάρια είναι το πακέτο. Και τώρα διάφορες χώρες ζητούν διαφορετικά πράγματα από το Πράσινο Ταμείο. Το οικονομικό πακέτο λοιπόν θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διασφαλίσει τη στήριξη των στόχων μας στο μέλλον. Με ρωτάτε επίσης πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της υλοτομίας και της αποψήλωσης. Κοιτάξτε, υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχει βιομάζα και προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση της βιομάζας και στο σύστημα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα, αλλά να μην αυξηθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τύποι βιομάζας που να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάντως είναι να χρησιμοποιήσουμε τους λιγότερο επιθετικούς τρόπους ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά συγχρόνως να βοηθήσουμε τις υπονάπτυξη χώρες να πετύχουν τους στόχους που θέλουμε να θέσουμε και να έχουν τη στήριξή μας γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χωρίστη Αμπαούντς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Κανιέτε. Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι σαφές. Αν μας αναφέρετε αυτές, ουσιαστικά αποφεύγετε τα πραγματικά θέματα. Δεν μιλάω σαν οικολόγος απαραίτητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω για την υδρορογμάτωση. Για να αποφασίσετε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία από αυτού θα λάβετε υπόψη σας την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών κατά της δρομάτωσης. Δεύτερον, εκ μέρους Μπενέγα και της Αστούρ, που θυμούνται πολύ καλά πώς αντιμετωπίσατε εσείς την καταστροφή του Πρεστίζ. Πώς θα φροντίσετε να πιέσετε την Ισπανική κυβέρνηση για να αποφύγει τη χρήση υδροκιανίου στις διάφορες διαδικασίες παραγωγής. Απάντηση το Ισπανικό κράτο πρέπει να τηρήσει όλε τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ όπω και οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δικιά μου υποχρέωση ω επίτροπο είναι ακριβώ να φροντίζω να τηρούνται οι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Δεύτερον, επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο και στο πρεστή, το ατύχημα του πρεστή. Είπατε ότι ήταν καταστροφική αντιμετώπιση μου. Τότε ήμουν υπουργό Αλία. Και τι έκανα, έκλεισα τον χώρο που ψαρεύαμε εκεί στην Ισπανία, ώστε ακριβώς να προστατεύσω την υγεία των ε, πολιτών. Για μένα αυτό ήταν το πρώτο, η υγεία των πολιτών. Και στη συνέχεια βοήθεια προς τους αλείς, ώστε οι αλείς να μην υποφέρουν από την καταστροφή αυτή και να μπορούν από την αρχή μέχρι το τέλος ε, να αποφύγουν τη ζημιά στα διάφορα ληφτικά πεδία. Σας καλώ λοιπόν, όποιος θέλει, ας πάει στην Ισπανία, στη Βόρεια Ισπανία, και δείτε πόσο καθαρές είναι οι ακτές εκεί. Αυτό έκανα τότε για το Πρεστής, καθάρισα και τις ακτές. Και όσον αφορά τώρα την υδρορογμάτωση. Κάθε χώρα μέλος είναι κυρίαρχη να πάρει τις αποφάσεις της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε υποχρεώνει τις χώρες μέλη να αναπτύξουν την τεχνολογία υδρορογμάτωσης, ούτε τους υποχρεώνει ούτε τους απαγορεύει. Απλώς πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Αν αποφασίσουν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν την τεχνική υδρορογμάτωση, είναι υποχρεωμένε οι χώρε να έχουν την κατάλληλη τεχνολογία. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθεί να έχει όλα τα επιστημονικά στοιχεία που υπάρχουν, να έχει πραγματογνωμοσύνη και από την Ευρώπη αλλά και εκτό Ευρώπη, ώστε να φροντίσει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την υδρορογμάτωση σε συνεργασία με εσά και με το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα κάνει προτάσεις έχοντας συζητήσει με όλα τα διαφερόμενα μέρη και εσείς εκπροσωπείτε τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο Σάλφος Μαραγάλ, κύριε Αρίς μιλήσατε για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής σας ε, σε εταιρείε ε, πετρελαϊκές, αλλά όχι για κάτι άλλο βαθύτερο αυτά που κάνατε σε φορολογικούς παραδείσους. Ίσως να είναι νόμιμα αυτά, αλλά είναι απαράδεκτα από πλευράς ευρωπαϊκής ηθικής. Θεωρώ ότι είναι ασύμβατο να αναλάβετε τις ε, αρμοδιότητες που προτείνετε να αναλάβετε με αυτά που έχετε κάνει στο παρελθόν. Σέβομαι τις απόψεις σας. Δεν ε, συμφωνώ με τον νόμο για τις ακτές ή για τον εύρο που κάνατε. Όλα αυτά από πλευράς περιβάλλοντος ε, δεν είναι σωστά. Και νομίζω ότι αυτά που κάνουν τόσοι επιχειρηματίες είναι γνωστά. Σας ερωτώ, θα ε, συνεχίσετε εσείς η οικογένειά σας να έχετε οικονομικά ενδιαφέροντες επιχειρήσεις στις Αντίλες ή τον Παναμά και θεωρείτε ναι ή όχι ότι θα ήταν σκόπιμο να παρετηθείτε γιατί έτσι πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάνετε λόγω αυτών των πληροφοριών που λάβαμε. Θα σας απαντήσω με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο. Εγώ ποτέ δεν είχα οικονομικές δραστηριότητες σε εταιρείε που να είναι σε φορολογικούς παραδείσους. Ούτε έχω ε, οικονομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που να είναι σκοτεινές. Όλα όσα έχω κάνει τα έχω δηλώσει πάντα στις ισπανικές φορολογικές αρχές. όλα μου τα οικονομικά συμφέροντα είναι όλα δηλωμένα στην εφορία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν έχω μετοχές σε καμία εταιρεία στο εξωτερικό. Είχα κάποιες μετοχές και τις πόλησα ε, πώλησα διότι ήθελα να είμαι σε κατάσταση απόλυτης διαφάνειας. Και νομίζω ότι κι αν ήξερε ο πρόεδρος Γιούνκερ ότι είχα ακόμη αυτές τις ε, ε, μετοχές θα με είχε προτείνει. Εγώ τις είχα και τώρα τις πούλησα. Δεν έκρυψα ποτέ τίποτα. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι έχω απόλυτα ήσυχη απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή μου γιατί πάντα πλήρωνα τους φόρους μου ως πολίτης και είμαι πολύ ικανοποιημένο και πολύ ήσυχος γιατί πάντα το έπραξα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα ο κύριος Ταμπουράνο. Κύριε Κανιέτα, μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ασχοληθεί στην ουσία με τους ε, καταναλωτές που είναι πολύ σημαντικοί στον τομέα της ενέργειας και για το τι εκπομπές θα έχουμε. Σύμφωνα με μελέτες του ΟΣΑ, καταλάβαμε ήδη το 2008 ότι 80% των αποφάσεων για την ενέργεια από τους καταναλωτές λαμβάνονται από τις γυναίκες. Οι γυναίκες που είναι εκείνες που επίσης χρησιμοποιούν περισσότερο ε, τις δημόσιες συγκοινωνίες. Θα σταματήσετε λοιπόν τις διακρίσεις ε, τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες. Θα διαμορφώσετε μια πολιτική στον τομέα της ενέργειας που να λαμβάνει υπόψη τις επιλογές των γυναικών. Είστε διατεθειμένος να υιοθετήσετε μια προσέγγιση ίσης αντιμετώπισης έναντι των ε, γυναικών, για παράδειγμα, επιτρόπων. Έναντι όλων των γυναικών που θα συζητήσετε, με τις οποίες, για παράδειγμα, θα συζητήσετε στα πλαίσια των ε, ε, επαφών με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδη πυλώνα για μια δημιουργία, για μια Ευρώπη απόλυτα καλύτερη χωρί αποκλεισμού. Πιστεύω απόλυτα στην ισότητα ανδρών και γυναικών. Και από τότε που έχω αρμόδι... υπεύθυνε θέσει στην πολιτική, πολλοί Ισπανοί ευρωβουλευτέ το ξέρουν, πάντα ε, έδωσα στι γυναίκε θέσει ε, μεγάλη υπευθυνότητα. Τη μέγιστη ε, υπευθυνότητα η κυρία Φράγα για παράδειγμα τη έδωσα τη θέση για την αλληλεία την πιο σημαντική για την γεωργία και η υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή έχει επικεφαλής μια γυναίκα και η υπηρεσία για τις μελέτες περιβαλλοντικών πτώσεων έχουν επικεφαλής γυναίκα. Έχω πλήρη συνείδηση το πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να λαμβάνουν θέσεις λήψη αποφάσεων και πάντα το έκανα αυτό σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία και μπορείτε να το ελέγξετε τούτων ευθέντων. Έχω διαβάσει χθε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξέρω ότι έχει επίπτωση η κλιματική αλλαγή στις γυναίκες. Ε, αναφέρθηκαν πολλά. Και επίσης αναφέρθηκε ότι πρέπει να είναι γυναίκες στις σημαντικές θέσεις όταν θα λαμβάνονται αποφάσεις για την κλιματική αλλαγή. Διότι ακριβώς ε, όταν μιλούσαμε για την έκθεση για τις επιπτώσεις ε, της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία της Αφρικής είδαμε τι επιπτώσεις έχει στις γυναίκες, άρα οι γυναίκες πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρουν οι ε, απόψεις των γυναικών για τη διαμόρφωση των αποφάσεων. Και στο ιδιαίτερο γραφείο μου φυσικά θα υπάρχουν ίσως αριθμός ανδρών και γυναικών και επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου μου θα είναι γυναίκα και θα επιδιώξω η ισότητα των δύο φίλων να είναι πραγματικότητα και στις γενικές διευθύνσεις που θα υπάρχονται σε μένα. Και αν ε, με τιμήσετε θα φροντίσω να είναι γυναίκα ή επαναλαμβάνω η επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου μου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτς. Όταν πρόκειται για θέματα πυρηνικής ενέργειας, τότε υπάρχουν ε, πολύ διαφορετικές απόψεις. Η πλειονότητα των ε, περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι κατά των πυρηνικών. Αλλά σημαντικοί Αμερικανοί ερευνητές κατέδειξαν ότι για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, τη θέρμανση του πλανήτη, ο, η παραγωγή ενέργειας από πυρηνικές πηγές είναι πολύ θετική. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι δεν παράγει ε, εκπομπές. Είναι καθαρή. Ε, οπότε ρεαλιστικά ε, μέσω πρόθεσμα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε την ε, πυρηνική ενέργεια. Διότι το χαρτοφυλάκιό σας δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ενεργειακή πολιτική. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα ποιες είναι απόψεις για την πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ, όπως έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα, η απόφαση για την πηγή ενέργειας που θα αναπτύξει κάθε χώρα είναι θέμα της κάθε χώρας. Δεν είναι θέμα ότι ένας επίτροπος είναι περισσότερο υπέρ μιας ή άλλης πηγής ενέργειας. Ο επίτροπος έχει ως καθήκον να ρυθμίσει την παραγωγή αυτή. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει υπέρ μιας ενέργειας που είναι καθαρή, έτσι, όπως η πυρηνική, που έχει βέβαια το πρόβλημα των αποβλήτων, και γι' αυτό και εμείς έχουμε τις οδηγίες για τα πυρηνικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διασφαλίσει το ανώτατο επίπεδο προστασίας. Και αυτό ακριβώ είναι που έχουμε κάνει με τις οδηγίες για την πυρηνική ασφάλεια και με τις οδηγίες μας για τα απόβλητα. Δουλεύουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, συνεργαζόμαστε με την Euratom και διασφαλίζουμε ότι αν υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να αναπτύξουν την πυρηνική ενέργεια, μπορούν να το κάνουν εφόσον διασφαλίζουν προστασία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά που υπάρχουν προγράμματα από τις χώρες μέλη τα μελετούν και κοιτούν ποιοι μπορεί να είναι οι περιορισμοί σε αυτά. Από εκεί και πέρα οι χώρες μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια πηγή ενέργεια θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ε, στοιχηματίζουν στην πυρηνική ενέργεια, άλλες τις καταργούν όπως η Γερμανία και το Βέλγιο και άλλες θέλουν να φτιάξουν νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες, νέα, νέες τέτοιες μονάδες όπως η Ουγγαρία για παράδειγμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε οι διαδικασίες ε, ε, κατάργησης των πυρηνικών μονάδων γίνονται βάσει συγκεκριμένων κανόνων και ότι τα απόβλητα πηγαίνουν στους χώρους που προβλέπεται για αυτά και όταν υπάρχουν νέες πυρηνικές μονάδες αυτές να χτίζονται βάσει των πιο σύγχρονων προδιαγραφών για να διασφαλίσουμε προστασία από την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη. Τώρα θα περάσω την Προεδρία στο συνάδελφο Μπούζεκ, ο οποίος θα αναλάβει το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας, της ακρόασης αυτής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Τζοβάνι. Έχουμε περάσει από τη μία πολιτική ομάδα στην άλλη. Περνάμε στον επόμενο γύρο. Ο συνάδελφος Ιβο Μπελέτ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, εδώ είμαι μπροστά σας. Εκτιμώ πάρα πολύ την δέσμευση που αναλαμβάνεται απαντός ε, στον κύριο Κρότε όσον αφορά την μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ξέρετε ότι είμαστε σύμμαχοι στον ε, τομέα αυτό και ξέρετε πόσο πολύ μας ενδιαφέρει και το θέμα του backloading. Έχω όμως μια επιπλέον ερώτηση όσον αφορά αυτό το σημείο. Πώς θα συνδυάσουμε τις φιλοδοξίες αυτές με την απόλυτα θεμητή ανησυχία της βιομηχανίας. Και ιδιαίτερα τι εγγύσεις μπορείτε να δώσετε εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, σε αυτούς που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, και το τονίζω αυτό, καλύτερες επιδόσεις στη βιομηχανία, προκειμένου να καταπολεμηθεί η λεγόμενη διαρροή διοξιδίου του άνθρακα και ιδιαίτερα μετά το 2020. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε την πιο μεγάλη αγορά φρέκα στον κόσμο. Και αναπτύσσουμε τέτοιες αγορές και αναπτύσσονται κι αλλού, Οι Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε παραδειγματίζονται από αυτήν. Η Ελβετία. Στο μέλλον, μάλιστα, οι δικές μας αγορές θα πρέπει να συνδεθούν με τις υπόλοιπες στον κόσμο. Γι' αυτό και η ευθύνη που επομιζόμαστε είναι τεράστια για το πώς θα διαχειριστούμε αυτό το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά να έχουμε η υπόψη μας και τα συμφέροντα της βιομηχανίας μας γιατί μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά που πρέπει να φροντίσουμε. Και για να τα φροντίσουμε πρέπει να έχουμε ένα βιομηχανικό τομέα με σημαντικό μέρος στην οικονομία μας που να είναι ανταγωνιστικός. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να συνεχίσουμε με το σύστημα αυτό δωρεάν ε, παραχώρησης δικαιωμάτων για να αποφύγουμε ακριβώς τη διαρροή διοξιδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο που είχαμε μέχρι τώρα από τις μελέτες της Επιτροπής διαπιστώσαμε ότι δεν μεταφέρθηκαν επιχειρήσεις αλλού, δεν μετεκαταστάθηκαν εξαιτίας της αύξησης της τιμής άνθρακα. Μπορεί να αυξηθεί λίγο η τιμή. Τότε πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας. Συνεπώς, στους πιο αποτελεσματικούς θα δώσουμε δωρεάν δικαιώματα. Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα νέο σύστημα βέβαια, αλλά να λάβουμε υπόψη μας το πρόβλημα ορισμένων χωρών, οι οποίες εξαρτώνται πάρα πολύ από τον άνθρακα για τις δικές τους εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού και να δούμε τι εξαιρέσεις μπορούμε να προβλέψουμε για αυτές τις χώρες. Ώστε να στηρίξουμε τη... τον ηλεκτρισμό, τη βιομηχανία ηλεκτρισμού σε αυτές τις χώρες και παραγωγή ενέργεια γενικότερα. Έχουμε τεράστια ευθύνη, όντω όμω, να ανταμείψουμε αυτού που έχουν τι καλύτερε επιδόσει. Ευχαριστώ, κυρία Γκαρσία Πέρε. Ευχαριστώ. Κύριε Αρίας Κανιέτα, υποψήφιος επίτροπος για τις κλιματικές αλλαγές, για την κλιματική δράση, ήσασταν υπουργός μιας κυβέρνησης που ενέκρινε την νομοθεσία για τις ακτές που ήταν όνειδος για ολόκληρη την Ευρώπη και θα ισοπεδώσει το, την, την φυσική μας κληρονομιά. Εσείς ως αρμόδιος υπουργός ήσασταν κατά των δεσμευτικών στόχων για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Τώρα βέβαια μας λέτε ότι θα στηρίξετε τέτοιους δεσμευτικούς στόχους πέραν του χαρτοφυλακίου σας παραδεχτείτε ότι δεν μας κάνετε και τη ζωή εύκολη με κάποιες παράπλευες πληροφορίες. Προσβάλλετε όλες τις γυναίκες. Επίσης, για να συγκαλύψετε μια σαφέστατη σύγκρουση συμφερόντων, πουλάτε άρον-άρον τις μετοχές σας. Και μία μέρα πριν την ακρόαση, μόλις χθες, δηλώσατε ότι είχατε λάβει αμοιβέ από το Λαϊκό Κόμμα ενώ είχατε αποκρύψει εδώ και τρει μήνε την πληροφορία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δήλωση του πόθεν έσχε σα. ότι έχετε το ηθικό παράστημα για να γίνετε επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Ευρωβουλευτή. Έχω δύο σχόλια να κάνω. Εγώ ανέκαθεν και ως Υπουργός Περιβάλλοντος ψήφισε υπέρ των προτάσεων της Επιτρόπου Κόνι Χέλεγκαρτ και μπορείτε να δείτε τα πρακτικά του Συμβουλίου. Ήμουν ανέκαθεν στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπερψήφισα τις προτάσεις της. Ανήκα στην ομάδα για την πράσινη ανάπτυξη. Οι 13 ε, υπουργοί που ταχθήκαμε υπέρ των καθαρών ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και κατά των ορυκτών, ήμασταν εμείς. κατά των ορεικτών καυσίμων. Και τότε δεν ήμουν επίτροπος για καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πούλησα τις ε, μετοχές μου, οχι αρονάρον όπως είπατε, αλλά όταν έμαθα ότι με πρότειναν για Ευρωπαίο Επίτροπο. Με βάση τη διαφάνεια και τη συνέπεια. Και θέσπισα το νόμο για τις ακτές για να προασπίσω τα συμφέροντα πολλών Ευρωπαίων πολιτών που είχαν επενδύσει στην Ισπανία, είχαν αγοράσει κόπεδα στις Ισπανικές ακτές και μία ωραία πρωία τους λέει ένας νόμος ότι θα χάσουν την ιδιοκτησία τους. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανα για να προστατεύσω τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό το έκανα. Και δεν έχω αποκρύψει τίποτα. Τίποτα δεν έχω αποκρύψει, κυρία Ευρωβουλευτή. Στο βιογραφικό μου αναφέρεται ότι διατέλεσα πρόεδρος της ε, Εκλογικής Επιτροπής. Είναι πολιτικό αξίωμα και μάλιστα δεν αμοιβόμουν γι' αυτό. Απλώς είχα έξοδα παράστασης. Και μάλιστα από την πρώτη στιγμή περιέλαβα αυτό το στοιχείο στη δήλωση πόθεν έσχες και στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων προς την Επιτροπή από την πρώτη μέρα για να το γνωρίσει, να το αναλύσει και να το εγκρίνει η νομική υπηρεσία. Το δήλωσε και στην Ισπανική εφορία. Πλήρωσα τους φόρους μου. Ήταν απόλυτα διαφανής όλες μου οι δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφια επίτροπε για τη δήλωσή σας. Ο κύριος Άσλι Φόξ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κύριε κανιέτρη. Εδώ είμαι. Θα μάθετε ότι δεν ενδιαφέρομαι για το τι κάνει ο κουνιάδος σας, ε, πώς βγάζει το ψωμί του. Υπάρχουν 248 σχέδια κοινού συμφέροντος ε, στα πλαίσια του τμήματος 10 της ε, δυνατότητας συνδέοντας την Ευρώπη. 5,8 δις ε, εκατομμύριο προπολογισμό τους για 5 χρόνια. 7 χρόνια, συγγνώμη. Τα περισσότερα λοιπόν δεν θα χρηματοδοτηθούν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσετε για να αποφασίσετε ποια από αυτά τα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν και ποια όχι. Ίσως ο πρόεδρος θα μπορούσε να παρακαλέσει τους σοσιαλιστές να σταματήσουν να συζητούν με τους συμβούλους τους. Επιπλέον, επιπλέον πολλά λέγονται για προγράμματα για να βελτιωθούν η αγωγή φυσικού αερίου. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να βελτιωθεί και το ε, πλέγμα μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος στις χώρες μας. Θεωρώ ότι όλα τα προγράμματα της δυνατότητα, που δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθεί η Ευρώπη και να υπάρξουν διασυνδέσεις ως απόλυτη προτεραιότητα. Είναι αλήθεια ότι το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη έχει μόνο 5,8 δις. Ένα από αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι όταν θα έχουμε την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου θα προτείνω ότι θα πρέπει αυτό να είναι προτεραιότητα της Ένωσης και στο πακέτο για τα 300 δις ε, που θα εφαρμόσουμε θα επιδιώξω να υπάρξει χρηματοδότηση για αυτά τα προγράμματα και επιπλέον όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε να λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στην επιλογή των προγραμμάτων ε, ενωσιακού συμφέροντος κάναμε κάτι που είναι σημαντικό. Δεν αποφασίζει η Επιτροπή τι πρόγραμμα θα προωθηθεί. Έχουμε περιφερειακές ομάδες με τις ρυθμιστικές αρχές, ε, τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, διάφορα, το λειτουργούν το ε, ενεργειακό πλαίσιο και διάφορους άλλους φορείς εμπλεκόμενους για να εκτιμήσουν ποια είναι τα καλύτερα. Και για μένα τα καλύτερα είναι αυτά που βοηθούν την διασύνδεση χωρών, ούτως ώστε να αυξήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης. Αυτά τα προγράμματα θα προωθήσουμε. Αλλά θα το αποφασίσουν οι περιφερειακές ομάδες. Πρέπει να ε, επαφιέμεθα στα περιφερειακά όργανα, όχι να αποφασίζει για αυτά τα, προγράμματα, τα προγράμματα ε, ενωσιακού συμφέροντο η Επιτροπή, αλλά είναι περιορισμένη η χρηματοδότηση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και κατά την αναθεώρηση των προοπτικών θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερη χρηματοδότηση, γιατί αυτά τα προγράμματα αξίζουν στήριξη. Ευχαριστώ πολύ ο, η, ο κύριος Χιράουτα Βιδάλ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στήριξαν ε, πάρα πολύ την ε, διασύνδεση σε 10% στην Ευρώπη για τον ηλεκτρισμό και μάλιστα είπαν ότι για το 2030 θέλουν να είναι 15%. Η τήρηση του στόχου αυτού είναι το εμπόδιο για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης και μας δυσκολεύει επίσης να πετύχουμε τους στόχους μας ακόμα και για το 2020. Κάποιες χώρες μελή στις προσπάθειες που κάνουν για να πετύχουν τους στόχους αυτούς ανέπτυξαν τις ε, ανανεώσιμε πηγές ε, ενέργειας σε ένα βαθμό, χωρίς όμως να μπορέσουν να εξάγουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη το πλεόνασμα ενέργειας που είχαν. Τι θα κάνετε λοιπόν για να συνδέσετε τους στόχους αυτούς με τη, τους υπόλοιπους στόχους της κλιματικής ε, ατζέντα για να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο. Τι θα κάνετε με τις διασυνδέσεις αυτές και τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για να αυξήσετε την διασύνδεση ακριβώς αυτήν. Απάντηση. Μία από τις προτεραιότητες μου θα είναι προσωπικά να δώσω όθηση σε όλα τα προγράμματα διασύνδεσης που είναι τόσο ανάγκη στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Βαλτική και τελειώνοντας με την ε, Ιγρική Χερσόνησο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα προγράμματα αυτά για το μέλλον. Αλλά για να έρθω στη συγκεκριμένη ερώτησή σας όσον αφορά την Ιβηρική, είναι αλήθεια ότι είμαστε ένας ενεργειακός θύλακας. Ότι έχουμε αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές, αλλά με δύο προβλήματα τα δίκτυά μας δεν είναι αρκετά αφή ώστε να απορροφήσουν το πλεόνασμα που κατά καιρού υπάρχει και από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να εξάγουμε. Παρόλο που έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Πορτογαλία, ναι, στην Πορτογαλία ναι, αλλά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να εξάγουμε. Ούτε στις γειτονικέ ε, χώρες, Ιταλία, Ενωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι, ενώ αν είχαμε καλή διασύνδεση θα μπορούσαμε. Έχουμε κάνει κάποια βήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως προωθεί τον διάλογο ανάμεσα στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, ακριβώς ώστε τα προγράμματα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Και όπως λέει και η κυρία Δεκαστήγιο, υπάρχει και ένα που έχει προχωρήσει κάπως περισσότερο. Μια διασύνδεση που περνάει από τα 400 στα 800 ΜΒ ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Τα άλλα καθυστερούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει πρώτα να πετύχει την πολιτική συμφωνία μεταξύ χωρών μελών ώστε να γίνει βιώσιμη η προσπάθεια αυτή και δεύτερον να βρεθεί η οικονομική στήριξη ώστε που είναι αναγκαία έτσι, για το ιδιωτικό τομέα ε, θέλει να έχει κάποιες εγγυήσει για να προχωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω από την άλλη θέλει και αυτή τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Θέλουμε λοιπόν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε όλες οι άδειες να δίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα. Θα αφοσιωθώ σε όλα αυτά και όχι μόνο για την Ιβηρική Χερσόνησο αλλά και για τις διασυνδέσεις ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριος Μύροσλαβ Ράνστορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, στον ενεργειακό τομέα έχουμε κάποια φυσικά μονοπόλια αλλά το μέλλον της ενέργειας στην Ευρώπη ε, θα προβλέπει μια καλύτερη αξιοποίηση και ένα συνδυασμό των μεγάλων και των μικρότερων ενεργειακών δομών και υποδομών. Πώς θα εξισορροπήσουμε τις ε, μεγάλες με τις μικρότερες ενεργειακές δομές. Απάντηση. Πιστεύω ότι για να βρούμε την ισορροπία θα πρέπει καταρχήν να πατάξουμε τις μονοπωλιακές πρακτικές. Αν υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, θα θέσω το ζήτημα στον αρμόδιο επίτροπο ανταγωνισμού για να διορθώσουμε τις περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας όμως είναι μία εσωτερική αγορά με τερματικούς σταθμούς. Δηλαδή, στο τρίτο ενεργειακό πακέτο θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως όλα τα στοιχεία. Και φυσικά χρειαζόμαστε και νέα μέτρα για τα ευφύη δίκτυα, για τις διασυνδέσεις, για τις διασυνοριακές μεταφορές και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, γιατί θα πρέπει να δέσουμε τον καταναλωτή στο επίκεντρο του ενεργειακού συστήματος. Θέλουμε έξυπνους μετρητές, θέλουμε αποδοτικές οικιακές συσκευές με οικολογικό σχεδιασμό. Να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν τις καλύτερες ενεργειακές επιλογές. Θέλουμε ευφύ ενεργειακά δίκτυα, συμπερίληψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και φυσικά πρόθεση της αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής. Όλα αυτά θα τα επιτύχουμε και μια αρμονική σύνυπαρξη μεταξύ των διαφόρων στοιχείων με μια ολοκληρωμένη και διαφανή εσωτερική αγορά της ενέργειας. Είπα στην αρχή ότι βασικός μου στόχος είναι η συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Και θα ήθελα κατά το τέλος της να έχουμε μια εύρυθμη εσωτερική αγορά με διαφανή και οριζόντιο υπολογισμό των τιμών. Γιατί αν έχουμε μια ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά θα ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε και μεγαλύτερη σύγκληση των τιμών προς τα κάτω. Αν συνεχίσουμε με κατακαιρματισμό τη αγοράς και απομονωμένε αγορές, ούτε ανταγωνιστικότητα θα έχουμε, ούτε ε, υγιή ανταγωνισμό, ούτε χαμηλέ ενεργειακέ τιμέ. Ευχαριστώ. Κύριο Κλώτ Τούρμε. Κύριε Κανιέτε, ως Ισπανός ε, Υπουργό Περιβάλλοντο, περιβάλλοντο, σα υπέρ τη ε, ε, υπέρ τη ε, εισαγωγή ε, βρώμικων άμμων από τον Καναδά και επίσης θελήσατε τα παλιά πυρνικά εργοστάσια να συνεχίσουν να λειτουργούν. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνούσατε ή ήσασταν υπερβολικά αδύναμος για να παρεμποδίσετε. Τώρα, ο Μιγγέλ Ντομέξολης δεν είναι κάποιος δεν είναι κάποιος ε, κουνιάδος σας. Είναι εδώ και 25 χρόνια μέλος της οικογένειάς σας αλλά και ε, ε, συνεταίρος σας επιχειρήσεις. Και επίσης εδώ και 13 χρόνια υπάρχει μια διαδικασία φόρο διαφυγής για μια επιχείρηση στην οποία παίζατε κύριο ρόλο. Πώς θέλετε με τέτοια δαμόκλειο πάθη από πάνω σας να αναλάβετε τέτοια ευθύνη. κύριε Τούρμες. Δεν ξέρω πού τις έχετε αυτές τις πληροφορίες. Κοιτάξτε. Στην δήλωση συμφερόντων μου υπόθηκε ότι η... αναφέρεται ότι εγώ είμαι δικηγόρος. Έχω λοιπόν ε, διατελέσει σύμβουλο σε πολλές πανικές εταιρείες. Και ως Υπουργός Περιβάλλοντος δεν έλαβα τις αποφάσεις αυτές. Στις κυβερνήσεις περνά η άποψη κάποιου υπουργού κάποιε φορέ και άλλε όχι, όπω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ μπορεί να κέρδισα όσον αφορά το backloading, αλλά έχασα άλλε μάχε, Αλλά τι μάχε πρέπει να τι δίνει κανεί. Ήμουν υπουργό περιβάλλοντο και επέβαλα μελέτε επιπτώσεων για όλα τα προγράμματα και μάλιστα τι πιο αυστηρέ που ποτέ υπήρξαν στην Ισπανία με, κριτήρι, με κριτέ, κριτήρια πάντα, πάντα παραλαμβάνω επιστημονικά και τεχνικά, όχι πολιτικά. Και αναφέρεστε τώρα σε αυτά, αυτές τις άμμους πίσας. Και υπάρχει και το θέμα των βιοκαυσίμων εδώ. Και το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει κυρίαρχα τι θα γίνουν αυτά τα θέματα. Όταν θα υπάρξουν ε, κοινοτικές ρυθμίσεις που επιτρέπει να γίνεται κάτι, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να αντιπαρατεθεί. Η Ισπανία συμμορφούται με την Ισπανική νομοθεσία και αν δεν το κάνει θα υπάρξουν δράσεις και προσφυγές της ε, Επιτροπής ε, εναντίον της. Εγώ ως Επίτροπος θα σεβαστώ αυτήν την ε, νομοθεσία. Εάν γίνει πιο αυστηρή η κοινοτική νομοθεσία και απαγορευτεί η εισαγωγή άμων πίσας όπως συζητιέται αυτή τη στιγμή στον ΠΟΕ τότε θα ε, το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή στην οδηγία για τα βιοκαύσιμα δεν γίνονται αυτές οι διακρίσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος David Coburn. Υποψήφια Επίτροπε, σαν ε, ένας ε, άντρας που γίνεται όλο και πιο διάσημος μιλώντας για τις πνευματικές ικανότητες των γυναικών, εγώ θα σας ρωτήσω για την ρήπανση και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλάει για την μείωση 40% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα όταν εκπέμπουμε 12% και το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 2%. Δεν συμφωνείτε ότι με τον τρόπο αυτό θα ξοδευτούν φοβερά πολλά χρήματα για μέτρα μετριασμού της ε, ρήπανση που καταστρέφουν την οικονομία. Ενώ στην πραγματικότητα ό,τι και να κάνουμε τελικά για τις εκπομπές, οι εκπομπές θα αυξηθούν παγκοσμίω. Κάθε Κινέζος, κάθε Ινδός θέλει ένα ψυγείο, θέλει μια Φεράρι κτλ. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω και για την οικογένειά σας. Πάντως Διακόπτει το μικρόφωνο του ομιλητή ο πρόεδρος. Έληξε ο χρόνος σας, συνάδελφε, έληξε ο χρόνος σας. Παρακαλώ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, να απαντήσετε παρακαλώ. Πρώτον, Νομίζετε ότι δεν χρειάζονται μέτρα. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Αυξάνει η θερμοκρασία του πλανήτη μα. πρέπει να περιοριστεί αύξηση αυτή στους δύο βαθμού. Λέτε, γιατί να κάνουμε κάτι αφού εμεί ρηπαίνουμε κατά 11%. 40% μείωση των εκπομπών δεν έχει καμιά σχέση με το επίπεδο εκπομπών που έχουμε. Έχει να κάνει με την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε την ε, μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς. Και χρειάζεται κάποιος να έχει τον ηγετικό ρόλο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και αυτός που έχει αυτό τον ηγετικό ρόλο είμαστε εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κοπεχάγη και σε όλες τις διασκέψεις κορυφής που έγιναν για αυτό το θέμα. Και πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι το Παρίσι και να πείσουμε και άλλους να πάρουν τα ίδια μέτρα όπω παίρνουμε και εμεί, Γιατί δεν γίνεται να λέμε αφού δεν κάνουν οι άλλοι δεν κάνουμε ούτε και εμεί, Μα δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Η καταστροφή μα περιμένει αν δεν γίνει κάτι. Για να πείσουμε του κινέζου, οι Ηνωμένε Πολιτείε να προχωρήσουν με φιλόδοξου στόχους για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, πρέπει να έχουμε ηγετικό ρόλο και να βρούμε και τα μέσα, γιατί αν θέλουμε μια πράσινη οικονομία, τότε θα γίνουμε ανταγωνιστικοί τότε θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Τέσσερα εκατομμύρια είναι σήμερα στην πράσινη οικονομία. Και είναι ο τομέας όπου έχουν χαθεί λιγότερες θέσεις απασχόλησης, που έχει ε, διατηρηθεί το επίπεδο και μέχρι το 2030 με τους φιλόδοξους στόχους μας θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, εκατομμύρια. Αυτό είναι ο στόχο μα. η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητά μα στην πράσινη οικονομία. Οι χώρε σα είναι μια από τι πιο ανταγωνιστικέ στην πράσινη οικονομία, με νέα προϊόντα, νέε προδιαγραφέ. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι ο στόχο που πρέπει να πετύχουμε. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό. Αν πιστεύουμε στο περιβάλλον, πρέπει να πιστέψουμε και σε αυτού του στόχου. Ευχαριστούμε κύριε υποψήφια επιτροπέ. Ο κύριο Μάρκο Πίπερ είναι ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Κανιάτα που με τόσο διαφανή και πλήρη τρόπο δηλώσατε τα οικονομικά σας συμφέροντα και νομίζω ότι και η δήλωση ότι λυπάστε για αυτά που είπατε για θέματα ισότητας γυναικών έπεισαν τους συναδέλφους. Θέλω να πω κάτι για την ενεργειακή απόδοση. Πολλά κράτη-μέλη έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα να επιτύχουν τους στόχους εξοικονόμησης που τους τίθενται γιατί είναι πολύ αναλυτικοί και γιατί είναι και ιδιαίτερα γραφειοκρατικοί. Κύριε Κανιέτε, πώς θα μπορούσαμε περισσότερη ευελιξία και με περισσότερα κίντρα να φροντίσουμε κάθε χώρα να αξιοποιήσει τα προτερήματά της, για παράδειγμα για τις ανανεώσιμες και για τα θέματα μείωσης του διοξείδιου του άνθρακος, ούτως ώστε κάθε χώρα να μπορέσει να συμβάλλει επιτυχέστερα στη συνολική ε, εκπλήρωση των στόχων συνολικά της Ευρώπης. Ο κύριος Κανιάτα. Για να, για να επιτύχουμε τους γενικούς μας στόχους, πρέπει να γίνει σωστή κατανομή των στόχων ανά κράτος μέλος με ευφύ τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τι δυνατότητες έχει κάθε κράτος μέλος και την κατάστασή του. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να γίνει και για το σύστημα εμπορίας, όπου υπάρχει ένα σύστημα καθορισμού προδιαγραφών, benchmarking, για το πώς δίδεται στόχο σε κάθε εταιρεία, εταιρεία και Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση κάθε χώρας και τις ανανεώσιμες. Δεν θα είναι δεσμευτική πλήρως η στόχη, αλλά θέλουμε δεσμεύσεις από διάφορα κράτη-μέλη, οπότε υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας με βάση τι ευκαιρίες, αλλά και τι ουσιαστικά δυνατότητες με βάση την μορφολογία του έχει το κάθε κράτος μέλος. Γιατί κάποιες δυνατότητες μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτύξουν ανανεώσιμες και άλλες όχι. Αλλά θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον 27% ανανεώσιμες. Και για την ενεργειακή απόδοση έχουμε πολλές δυνατότητες. Γιατί μπορούμε να εργαστούμε ακόμη και σε επίπεδο του κάθε πολίτη. Μπορούμε να ε, κάνουμε τις μεγαλύτερες οικονομίες στον τομέα των οικοδομών και στον τομέα της θέρμανσης. Να βοηθήσουμε λοιπόν ακόμη και τον κάθε πολίτη να επιλέξει τη μορφή θέρμανσής του για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντικά μέσα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, πολύ σημαντική ε, οδηγία, με την απόδοση των κτηρίων και επίσης θέλουμε να έχουμε και ευφύς μετρητές όλα τα συστήματα. Εάν το επιτύχουμε θα έχουμε σε κάθε χώρα πολύ καλές εξοικονομίες ενέργειας, ε, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Μπορούμε να έχουμε 100 εκατομμύρια ευφυεί μετρητέ στο μέλλον στην Ένωση και αυτό θα επιτρέψει σε κάθε καταναλωτή να είναι αποτελεσματικός. Ευχαριστώ κυρία Καβεσόν Ρουίς. Ευχαριστώ. Κύριε Κανιέτε. Ε, τα λόγια έχουν μεγάλη δύναμη και σήμερα άκουσα πολλές υπερβολές που θα μπορούσα και να τις πιστέψω αν δεν είχα ήδη απείρα από την Ισπανία γιατί γνωρίζω τις πολιτικές σας και όντως σπεύσετε να διορθώσετε την δήλωση, ακόμη και όταν ήσασταν γερουσιαστής. Θα συλλητεύσετε την κυβέρνησή σας και θα ε, επιβάλλετε κυρώσεις ε, αν δεν, πληρώσει, δεν συμμορφωθούν τους στόχους του 2020. Εσείς καταστρέψετε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και με άδικο και ψευδό τρόπο μιλήσετε για ένα ε, έλλειμμα στο οποίο εσείς συμβάλλατε. Επίσης, ε, ε, θα δώσετε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για αυτοκατανάλωση και εκδημοκρατισμό της ενέργειας, ενώ για τα θέματα αυτά δημιουργήσατε πολλά εμπόδια στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ξεκινώντας από το, από το πρώτο θέμα που είπατε, στην Γερουσία ε, στην, και στην Ισπανική Βουλή δεν απέκρυψα κανένα στοιχείο. Όλα βγήκαν αυτά στον τύπο. Και τι έκανε η κυβέρνηση, τι ήταν ε, το περίεργο που έκανε. Δημιούργησε ένα έλλειμμα στις, ε, στην τιμολόγηση εξαιτία των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια υπερβολικό. Εσάς, εσείς δεν το θεωρείτε ίσω υπερβολικό, αλλά τελικά την ύφη την πληρώνουν οι καταναλωτέ. Και μάλιστα αυτό εξαιτία μια ασφαλμένης πολιτικής που οδήγησε σε έσοδα άνω του 20% που για σας μπορεί να είναι ε, σημαντικά, αλλά δεν είναι δεν... Ε, για σας μπορεί να είναι λογικά, αλλά δεν είναι λογικά για, το... για τα δημόσια οικονομικά. Ε, εμείς είμαστε υπέρ ε, μεγαλύτερης λειτουργίας της οικονομίας αγοράς και περιορισμού των κρατικών ενισχύσεων. Πάντως εγώ ως Επίτροπος θα εφαρμόσω την κοινοτική, την ενωσιακή νομοθεσία και θα επιβάλλω κυρώσεις και στην Ισπανική κυβέρνηση και σε οποιοδήποτε κράτος που θα παραβιάσει τους στόχους εφόσον είναι δεσμευτική. Αλλά μην ανησυχείτε, το 2013 η Ισπανία ήταν στο 16,1% και το 20% θα πάει στο 20%. Είναι από τις καλύτερες ε, ε, χώρες ε, με τις καλύτερες επιδόσεις στην ενέργεια. Δεν είναι ουραγός στην υλοποίηση των στόχων. Βέβαια, αν το 2020 δεν υλοποιηθούν οι στόχοι, θα πρέπει να εξετάσουμε τα αίτια της μη συμμόρφωσης. Επίσης, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι επιβάλλει κυρώσει, αλλά να βοηθάει για την εφαρμογή τη ερωσιακή νομοθεσία. Βέβαια, αν κάποιε χώρε την παραβιάσουν, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα υποστούν κυρώσει. Εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εκπροσωπώ την Ισπανία, αλλά το συμφέρον 500 εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Αυτό είναι το καθήκον μου, αυτή είναι η δέσμευσή μου και αυτό θα κάνω αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνκαν είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, γνωρίζετε ότι η Σκοτία παράγει ενέργεια, είναι σημαντικός παραγωγός και υδρογονοθράκων και ανανάσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζω να έρθετε στη Σκοτία και να δείτε από μόνο σας πώς έχει η κατάσταση εκεί. Άκουσα τη στήριξή σας για το αβόριο δίκτυο, πολύ καλό αυτό. Θα θέλω όμως ένα χρονοδιάγραμμα και να μας πείτε και οικονομικά τι θα προβλεφθεί. Όσον αφορά την υδρορογμάτωση τώρα, δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα ότι οι χώρες μέλη έχουν την αρμοδιότητα. Τι θα κάνετε όμως ώστε να εξακολουθήσουν να έχουν αρμοδιότητε οι χώρες μέλη για το ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά την ε, υδρογραμμάτωση μεταξύ άλλων, γιατί ξέροντας ότι και το φυσικό αέριο μπορεί να εμποδίσει την ε, μετακίνηση προς άλλες πηγές ενέργειας απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η Βόρεια Θάλασσα, η πρωτοβουλία για το δίκτυο αυτό, είναι κάτι βέβαια που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την διασύνδεση. Συνεπώς θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε να προσπαθήσω να δω πώς θα στηρίξουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και προγράμματα. Ξέρουμε ότι τα κονδύλια είναι περιορισμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει και με τη διασύνδεση στη Βαλτική. Θέλουμε και εκεί να βοηθήσουμε, γιατί όντω, όπω σα είπε, η διασύνδεση πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η περιφερειακή προσέγγιση έχει τεράστια σημασία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μία ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά. Μπορούμε όμω να αρχίσουμε να τη φτιάχνουμε από το περιφερειακό επίπεδο, από περιφερειακές ολοκληρωμένες αγορές που θα αναπτύξουμε και θα τις συνδέσουμε μεταξύ τους ώστε να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά τελικά που είναι και το τελικό αποτέλεσμα στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε. Υπάρχουν καλά παραδείγματα στις χώρες Μπενελούξ για παράδειγμα, που συμμετέχει και η Γερμανία. Υπάρχει αυτό το υπεράκτιο πλέγμα, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο την περιφερειακή προσέγγιση. Παντού, ώστε να διασυνδεθούν όχι μόνο οι είδη ενέργειας, για να λύσουμε όσο γίνεται καλύτερα το πρόβλημα αυτό της ενέργειας. Όσον αφορά τώρα το σχεστολιθικό αέριο θα μελετήσω πώς λειτουργεί το σύστημα και θα υιοθετήσω νομοθεσία εφόσον προηγουμένως έχουμε δει τι θα γίνει στην Ευρώπη με την αρχική εμπειρία που θα έχουμε. Χωσέ Ιγνάτσιο Γαρία τώρα. Κύριε Κανιέτε. Στην γραπτή σας απάντηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλήσατε για την ανάγκη όλοι οι τομείς μεταφοράς να συμβάλλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν πολλές ελλείψεις ε, και στις αερομεταφορές και στις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει να ελέγξουμε τις, ε, τα καυσαέρια της ναυτιλίας και μετά να περάσουμε στον περιορισμό. Αλλά μην ξεχνούμε και τις αερομεταφορές. Ε, η, μόλις, η ρήπαση του περιβάλλοντος από τους δύο τομείς ε, μεταφορών έχουν σημαντικές ε, επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Επίσης, οι διεθνείς αερομεταφορές έχουν εξαιρεθεί από το Διεθνές Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Σκοπεύετε να υιοθετήσετε πρωτοβουλίες πιο περιοριστικές και για τις θαλάσσιες μεταφορές και να μην δημιουργηθεί δυσμενής θέση της, ε, του ευρωπαϊκού κλάδου σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επίσης, τι θα γίνει με τους αερομεταφορές μετά το 2016. Θα, δεν θα πρέπει να περιληφθούν και τα καυσαέρια και αυτό το τομέα για να συμβάλλει και αυτός μέχρι το 2016 στον περιορισμό των καυσαερίων. Σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και όντως, αυτή τη στιγμή έχουμε διαφοροποιημένη συμμετοχή των διαφόρων τομέων. Στην περίπτωση των μεταφορών και δι των αερομεταφορών, εμπίπτει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών το ενδο, οι ενδοκινοτικές αερομεταφορές. Οι μεταφορές όμως ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα. Η ρύθμιση του προβλήματος αυτού θα πρέπει να λάβει υπόψη την ε, Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και το κατά πόσο θα μπορέσει αυτός ο οργανισμός να θεσπίσει μέτρα για την παγκόσμια αγορά. Αν το 2016 στην συνεδρίαση που θα γίνει στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας υποβληθούν θεσμευτικά μέτρα, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αν όμως δεν καρποφορήσει αυτή η συνεδρίαση και δεν θεσπιστούν κάποια παγκόσμια μέτρα, αν η Παγκόσμια Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας δεν τα καταφέρει να επιβάλλει δεσμευτικά μέτρα, τότε θα πρέπει να επανέλθουμε στην προηγούμενη οδηγία και θα πρέπει εμείς και εσείς να λάβω μία απόφαση για να δούμε αν θα την εφαρμόσουμε πλήρως, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, ή θα πρέπει να την τροποποιήσουμε. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το 2016 για να δούμε τις εξελίξεις στην αρμόδια οργάνωση που ρυθμίζει τις αερομεταφορές. Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός θα εγκύψει και αυτό στο θέμα αυτό. Εμείς ε, έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα ε, monitoring, ε, ενημέρωσης ε, και εξακρίβωση επαλήθευση για να δούμε ποιος ρηπαίνει. να δούμε αν κάποιος ρηπαίνει για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες, για να δούμε από πού προέρχονται οι εκπομπές στη, από την αυτιλία. Επίσης θα δούμε τι θα κάνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Αν δεν λάβει αποφάσεις, θα μπορούσαμε εμείς σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο να προτείνουμε κάποια μέτρα. Για τις δύο αυτές ε, μεταφορές, τις ναυτιλιακές και τις αερομεταφορές, περιμένουμε τους παγκόσμιους οργανισμούς να λάβουν κάποια μέτρα, γιατί είναι παγκόσμιο το θέμα και χρειάζεται μια παγκόσμια απάντηση. Κυρία Πιετικάινεν. είναι. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Με συγχωρείτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος αλλά κατάλαβα ότι δεσμεύεστε ιδιαιτέρως να καταπολεμήσετε την κλιματική αλλαγή που θεωρείτε ότι είναι πολύ σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα, ότι δεσμεύεστε να εργαστείτε για να υπάρξει αυτό το αποθεματικό για την ε, σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών και για άλλα μέτρα και θέλετε να υπάρχουν ευφιέστατα πανευρωπαϊκά δίκτυα, super smart, και επίσης να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις και επίσης περισσότερες ανανεώσιμες. Θα ήθελα όμως λίγο περισσότερα σχόλια για αυτά. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιούμε ε, τις ε, ε, ενεργειακούς πόρους τρομερά πολλούς και θα χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερους. Με συγχωρείτε κυρία μου. Κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα. Αναφέρατε ένα ποσό. Τι ποσό, δεν κατάλαβα. Μία πρόταση. Παρακαλώ. Η ερώτηση. Πώς θα βοηθήσετε να έχουμε περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλές ε, δυνατότητες για να έχουμε περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, οι ανανεώσιμες. Μπορούμε να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες και επίσης να βοηθήσουμε μέσω νέας έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανία να αξιοποιήσει περισσότερο τις ανανεώσιμες. Έχουμε για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά και την αιωλική ενέργεια. Υπάρχουν και άλλες μορφές ανανεώσιμες. Για παράδειγμα, υπάρχει η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και, αυτή την, ε, και αυτόν τον κλάδο μπορούμε να αναπτύξουμε άρα θα δημιουργώντας έτσι και ε, θέσεις εργασίας και μειώνοντας ε, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επίσης περισσότερη ενεργειακή απόδοση. Να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας στις κατασκευές. Να εργαστούμε μαζί με τον κλάδο για να το επιτύχουμε. Αυτή τη στιγμή ανανεώνουμε μόνο 1% των κτηρίων μας ε, των χρόνων. Αυτό είναι πολύ λίγο. Να περάσουμε στο 2. Αυτό δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, αυτό δημιουργεί πολλές πράσινες θέσεις εργασία. Επίσης να χρησιμοποιήσουμε διάφορες συσκευές που θα μειώσουν την παραγωγή ενέργειας. Έχουμε τον οικολογικό σχεδιασμό των συσκευών. Θα μπορούσε να βοηθήσει και την ε, ε, η οικολογική σήμανση των συσκευών. Μπορούμε να αναπτύξουμε πολλούς τομείς. Καλύτερες τεχνικές καύσεις, ε, καλύτερες εγκαταστάσεις ε, στην, στα εργοστάσια για καλύτερη καύση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε από την ενέργεια υψηλού άνθρακα στην ενέργεια χαμηλού. Η κυρία Σιμώνα Ποναφέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του κύριου Γιούγκερ, ακούσαμε για επιπλέον 300 δισεκατομμύρια επενδύσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς. Η Ευρώπη πρέπει όντως να επενδύσει και ε, στον τομέα για τον οποίο εσείς είσαστε αρμόδιος. Οπότε θέλω να σας ζητήσω να μου πείτε αυτά τα 300 δισεκατομμύρια πού θα χρησιμοποιηθούν όσον αφορά τις ενεργειακές αλλαγές και τη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης. Ποιε θα είναι οι προτεραιότητέ σα λοιπόν σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να ενθαρρύνουμε και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια αλλά και την ενεργειακή επάρκεια. Και τι θα γίνει με τα δίκτυα, πώς θα τα αναπτύξετε περισσότερο απάντηση. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία με αυτήν τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποφεληθούμε δηλαδή από επενδύσεις στον τομέα ε, της ενέργειας και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του κοινοτικού προϋπολογισμού, γιατί έχουμε ένα mainstreaming για όλα τα μέτρα, δηλαδή ώστε το 20% όλων των μέτρων να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση ανώσιμων πηγών αέρης κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει ότι οι χώρες μέλη θα χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνουν τα διαφορετικά ταμεία ώστε να κινητοποιήσουν πόρους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν που έχουμε από το πακέτο 2014-2020 είναι ότι τα πρώτα χρόνια 2014 καταρχήν, το ποσοστό χρήσης των κονδυλίων ε, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι της τάξης του 12%. Τώρα όταν αρχίσουν και οι εταιρικέ ε, συμφωνίες, ε, το greening κτλ, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε το 12%. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να βρει νέα συστήματα χρηματοδότησης προγραμμάτων, ομόλογα έργου και άλλες μορφές βοήθειας που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Και στο πακέτο αυτό των 300 δισεκατομμυρίων η ενέργεια, η ενεργειακή επάρκεια και ανανόσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε και υπό την ε, Αντιπρόεδρο για την Ενεργειακή Ένωση αλλά και με τους υπόλοιπους επιτρόπους με εκείνον για την απασχόληση για παράδειγμα να κινητοποιήσουμε πόρους υπέρ της ε, ενέργειας. Με τον πρόεδρο Γιούγκερ, λοιπόν, με τα διευθυντικά ταμεία, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούμε να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα υπέρ της πράσινης οικονομίας. ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάβιο Τζανανάτ. Α, συγγνώμη. Πρώτα ο κύριος Πολ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο εδώ στο Κοινοβούλιο μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε κάποιον που έχει εργαστεί στην πράξη γνωρίζει τα θέματα αυτά, μας φέρνει την εμπειρογνωμοσύνη. Είναι καλό να έχουμε τέτοιους που ήταν και στο Κοινοβούλιο τώρα σε επιτρόπους. Τι μέτρα θέλω να ρωτήσω μπορούμε να κάνουμε για την παραγωγή και για τους καταναλωτές. Πώς δηλαδή μπορούμε μέσω των καταναλωτών να έχουμε περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια ιδίω τα ιδιωτικά νοικοκυριά. Δηλαδή οι τιμές της ενέργειας να πέσουν γιατί ξέρετε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα ενεργειακής και πώς θεωρείτε ότι η αποκέντρωση της παροχής ενέργειας μπορεί να βοηθήσει. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι στα πλαίσια των ευφυών τεχνολογιών θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρέπει να αναπτύξουμε τα ευφυή δίκτυα και τους ευφυείς μετρητές. Είναι πολύ σημαντικό ο καταναλωτή να είναι στο κέντρο τη λήψη αποφάσεων. Πρέπει να μπορεί να επιλέξει πότε να καταναλώσει, πόσο να καταναλώσει, να γνωρίζει πάντα την ενημέρωση, αλλά με προστασία των δεδομένων. Πολύ σημαντικό, πολύ Επίσης, αν αποφασίσει ο καταναλωτής να παραγάγει τη δική του ενέργεια μέσω αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις γι' αυτό. Πρέπει να υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο. Θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για να υπάρχουν κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. Γιατί κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική προσέγγιση. Είναι ένα από τα θέματα για τα οποία έχει προστιθέμενη αξία η ευρωπαϊκή ρύθμιση. Πρέπει να ρυθμίσουμε πώς μπορεί να παραγάγει ενέργεια ο καταναλωτής, αλλά πώς θα συνδεθεί επίσης με το δίκτυο. Και μπορεί να χρειαστούν κάποιες επιδοτήσεις γι' αυτό και πώς θα ενταχθεί στο δίκτυο. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Πώς θα το κάνουμε. Και βεβαίως ε, υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που πάσχουν από ενεργειακή φτώχεια, που δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Έχουμε και συστάσεις ε, του Φόρουμ Πολιτών γι' αυτό. Ποια πρέπει να τα μέτρα, ποιος είναι ο ορισμός των ενεργειακά ευαλώτων ατόμων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από κράτος σε κράτος. Χρειάζεται κοινή προσέγγιση λοιπόν. Αλλά είναι σαφές ότι κάποια τμήματα του πληθυσμού έχουν μεγάλο πρόβλημα να πληρώσουν για ενέργεια και θα πρέπει να βρεθεί καλύτερος τρόπος να τους βοηθήσουμε. Μέσω επιδομάτων ή μέσω ε, επιδοτήσεων για τα νοικοκυριά είναι περίπλοκα θέματα. Αλλά ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να τα δούμε και να προτείνουμε κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κανιέτε. Ο κύριος Φλάβιο Τζανονάτο. Ευχαριστώ. Εγώ έχω κάπως διαφορετική ερώτηση από αυτές που ακούσαμε επανειλημμένως. Πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα και ελαστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και χαμηλότερο κόστος. Αυτή ήταν η υπόσχεση που ακούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Στην υδροελεκτρική ενέργεια, βασική πηγή του ενεργειακού μείγματος. Μία ενέργεια υδροελεκτρική ε, είναι παρούσα στην Ευρώπη πάνω από έναν αιώνα και αντιπροσωπεύει το 26% του συνόλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το 69% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Ευρώπη, τα συστήματα παραχώρησης υδροελεκτρικής ενέργειας διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Κάποιες χώρες όπως Ιταλία, η Ισπανία και άλλες προσπαθούν να επιβάλλουν μια απελευθέρωση του κλάδου. Δυστυχώς διακόπτει τον ομιλητή ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ένα από τα αποτελέσματα του τρίτου ενεργειακού πακέτου ήταν ότι έχουμε όλο και πιο ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές στα κράτη-μέλη. Επιπλέον, έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Βαίνουμε προς μία οδό ευρωπαϊκής ρυθμίσης μέσω των ενώσεων εθνικών ρυθμιστικών αρχών και χάρη στην καλύτερη δικτύωση των φορέων των δικτύων και καλύτερο συντονισμό. Οδεύουμε προς μία εναρμόνιση. Βέβαια, όντως, ακόμη δεν έχουμε παρόμοιες καταστάσεις παντού και, και για την υδροελεκτρική ενέργεια έχουμε αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα. Πριν τη θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας, την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της αποτελεσματικής νομοθεσίας. Σημερίζομαι την ανησυχία σας, αλλά θα πρέπει να αναλύσουμε αν θα επιφέρει προς τη θέμενη αξία μία πανευρωπαϊκή νομοθεσία ή απλώς θα επιτείνει τη γραφειοκρατία. Έχουμε αρμόδια αντιπρόεδρο που θα συντονίσει το το θέμα του εύνομοθετήν. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να θεσπίζουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία για να επιφέρουμε προστιθέμενη αξία και ε, πλεονεκτήματα που δεν μπορούν να επιφέρουν οι εθνικές νομοθεσίες. Ε, υπάρχουν βέβαια πολλά επιχειρήματα υπέρ της ολοκληρωμένης ε, εσωτερικής αγοράς, γιατί μια νέα αγορά, εσωτερική αγορά, θα έχει εναρμονισμένες τιμές, καλύτερη κυκλοφορία ενέργειας και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανταγωνισμό ε, θεμητό. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε, όπως είπα, τις αρχές αναλογικότητας και επικουρικότητας. Είναι σημαντικές για να ε, έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στο κύρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινωτικών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστούμε. Η κυρία Αγιούζο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, όπως μα είπε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και είναι η αρμόδια για να το πει. Εδώ δεν πρόκειται για την προσπάθεια μόνο της αριστερά, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει κόλλημα στη διαδικασία και επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια. Εσείς είσαστε αρμόδιος για να αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο που σας έχει προταθεί. Εδώ θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό είσαστε ακριβώ ο κατάλληλο άνθρωπο. Λοιπόν, σε σχέση με τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, φυσικό αέριο και τα προβλήματα που υπάρχουν σε διάφορε ευρωπαϊκές χώρες, εσείς πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική, η εξωτερική ενεργειακή πολιτική τη Ευρώπη τα επόμενα χρόνια και τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει στα εξωτερικά σύνορα και τι νέε διόδου μπορούμε να βρούμε, τι νέε διαδρομέ μπορούμε να βρούμε για την ενεργειακή μα κάλυψη. Απάντηση. Επιθυμία μου θα ήταν το South Stream, η διαδρομή αυτή, να αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί έτσι έχουμε μια απόλυτη εγγύηση ότι τηρείται η κοινοτική νομοθεσία. Αυτό είναι το επιθυμητό. Αλλά τον ε, νότιο διάδρομο πρέπει να τον προωθήσουμε και να φροντίσουμε ο ιδιωτικός τομέας να τον ενισχύσει. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε για τη διασύνδεση των βαλτικών χωρών, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, και να υπάρξει συγχρονισμός του ενεργειακού συστήματος ε, της Βαλτικής με το ευρωπαϊκό, κάτι το οποίο κοστίζει, αλλά είναι αναγκαίο γιατί διασφαλίζει ενεργειακή ανεξαρτησία. Πρέπει επίσης να βασιστούμε στις ε, ντόπιε πηγές ενέργειας, όσο γίνεται περισσότερο. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση, γιατί τότε θα αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε λιγότερο, θα εξαρτώμεθα λιγότερο από αυτούς που μας ε, εξάγουν φυσικό αέριο. Το ευρωπημένο αέριο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε να δημιουργηθούν hubs στη Νότια Ευρώπη. Πολλές δυνατότητες υπάρχουν συγχρόνως, αλλά να μην εξαρτώμεθα από μια ενιαία πηγή, από μια ενιαία πρόσβαση. Για τελείω θα δυσκολευτούμε από το φθινόπωρο. Όλοι μπορούμε να αγοράζουμε περισσότερο και πρέπει να ενωθούμε σε αυτό. Η Ευρώπη έχει μεγάλη αγοριστική δύναμη σε αυτό το τομέα στην ενέργεια και εγώ ως επίτροπος, εάν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φτιάξουν πλατφόρμες κοινέ για την αγορά ενέργειας και τηρούν τις ρυθμίσεις του ΠΟΕ και τους κανόνες ανταγωνισμού, τότε θα το στηρίξω. Η Ευρώπη μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ τη θέση της σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Η κυρία Γιούτε Ρούτελαντ. Κύριε Κανιέτε, το χαρτοφυλάκι όσος ε, λέγεται ότι πρέπει να είστε επικεφαλής των, προσπαθειών, των προσπαθειών για το κλίμα και τις ενέργειες για τις διαπραγματεύσεις. Μας αναφέρατε τους στόχους για τις εκπομπές, αλλά θέλουμε να μας μιλήσετε και για την ενεργειακή ασφάλεια. Θα προσπαθήσετε να υπάρχουν δεσμευτικοί φιλόδοξοι στόχοι για τα κράτη-μέλη, για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας και για ανανεώσιμες. συζητήσαμε επίσης και θέματα ναυτιλίας. Θα αγωνιστείτε ουσιοδός να σημειωθεί πρόοδος το θέμα αυτό γιατί η απάντησή σας ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που θα χαράξουν νέους δρόμους στον τομέα αυτό. Πολλές γυναίκες και κοπέλες θέλουν να μας πείτε επίσης τι πιστεύετε για τις διανοητικές τους, ικανότητες. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε για τα θέματα ναυτιλίας. Το θέμα με την ναυτιλιακή πολιτική είναι ότι πρέπει να ξέρουμε τι εκπομπές έχουμε πριν ε, προτείνουμε ανώτατα όρια ελέγχου μειώσεων. Πρέπει να ξέρουμε τι επίπεδο εκπομπών έχουμε. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει ένα ευφυές σύστημα παρακολούθησης υποβολής εκθέσεων για να δούμε ποιες είναι αυτές οι εκθέσεις και για να ελέγξουμε πόσες είναι. Μόλις έχουμε τα στοιχεία αυτά θα είμαστε σε θέση να λάβουμε αποφάσεις. Αλλά επειδή το πρόβλημα των ε, θαλασσίων μεταφορών είναι πλανητικό, διότι όπως ξέρετε τα μεγάλα πλοία ε, διασχίζουν τον κόσμο, πρέπει να υπάρχουν συνολικά μέτρα για τα πλοία από ε, κάποιες διαστάσεις και πάνω. Οπότε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, IMO, στην επόμενη συνάντησή του θα δει αν θα ληφθούν αποφάσεις για το θέμα αυτό ή όχι. Εάν δεν τις λάβει, θα τις λάβουμε εμείς. Διότι μας ενδιαφέρει τα πλοία μας να είναι αποτελεσματικά ενεργειακά και να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Δεύτερον, για τους στόχους ενεργειακής ε, ασφάλειας. Για την ασφάλεια, ασφάλεια της προμήθειας. Πρέπει να εργαστούμε σε όλα τα μέτωπα, ούτως ώστε όλες οι χώρες να έχουν εγγυημένη αυτή την ασφάλεια προμήθειας. Έχουμε το πρόβλημα με την Ουκρανία, γεωπολιτική σύραξη. Αλλά η αστάθεια μπορεί να υπάρξει, για παράδειγμα, στην Νότια Μεσόγειο. Μπορεί επίσης ε, σε άλλες συγκυρίες να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα πρέπει οι ροές να είναι αντιστρέψιμες, να έχουμε συστήματα, συστήματα διασύνδεσης με αντιστρέψιμες ροές και συστήματα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και αλληλεγγύης αναπεριοχές η ασφάλεια προμήθειας είναι πολύ σημαντική για μια Ευρώπη ανταγωνιστική στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χένα Βιρκούνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Κανιέτε. Όπως ξέρουμε, η συζήτηση αυτή τη στιγμή και η διαδικασία λήψη αποφάσεων για, τα για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές ε, έχει ε, χαράξει ένα σύνορο μεταξύ τους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στερεί επειδή δεν έχει μια γενική επισκόπηση κατάσταση. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την ενέργεια από το περιβάλλον. Θα πρέπει να φροντίσουμε για την ανταγωνιστικότητά μας και να εξασφαλίσουμε πρόσβαση ε, των επιχειρήσεων σε, προσιτή, σε ενέργεια σε προσιτές τιμές αλλά και φιλοπεριβαλλοντική. Ο πρόεδρος Γιούγκερ συνένωσε αυτά τα δύο θέματα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο για να διορθώσουμε το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει ε, το έργο της το Νοέμβριο. Κύριε Κανιέτε, ήδη μας είπατε πόσο σημαντική είναι η πράσινη φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ρωτώ λοιπόν ποια κατά τη γνώμη σα θα είναι τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν. δυστυχώ διακόπτει ο πρόεδρο στα μέσα της ερώτηση. Αν καταλάβατε κάτι απαντήστε, λέει ο πρόεδρος. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την εξασφάλιση της φιλοπεριβαλλοντικής ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης. Το πιο σημαντικό που θα πρέπει να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βεβαιότητα και ασφάλεια δικαίου. Μόνο με ασφάλεια δικαίου θα προσελκύσουμε επενδυτές για να επενδύσουν σε προγράμματα και σχέδια και σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Θα πρέπει να ξέρουν οι επενδυτές ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Και με το που θα συμφωνηθεί στο, τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο το πακέτο για το 2030 θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε συνεργασία με το περιβάλλον, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγγνώμη, συζήτηση για όλους τους κανόνες για να δούμε πώς θα αναπτύξουμε και θα μεταρρυθμίσουμε ε, την, το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών, την ε, οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, τι δεσμεύσει των κρατών μελών για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, το νέο σύστημα διακυβέρνησης και ούτω καθεξής, ώστε πολύ σύντομα να γνωρίζουν όλοι οι βασικοί μα εταίροι στον κόσμο ποιοι είναι οι κανόνε του παιχνιδιού. Επίση, οι, πολι... οι κλιματικές αλλαγές θα πρέπει οριζόντια να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές των διαρθρωτικών ταμείων. Και με τα κονδύλια που έχουμε προσημειώσει στο πακέτο Juncker θα μπούμε στο σωστό δρόμο για την πράσινη ανάπτυξη. Γιατί θα έχουμε επενδυτικέ ευκαιρίε σε πολλού τομεί. Ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά και στι διασυνδέσει. Θα υποβληθούν πολλά σχέδια και προγράμματα για τι διασυνδέσει. Έτσι θα εντατικοποιηθούν οι δραστηριότητε και θα γίνει πραγματικότητα η πράσινη ανάπτυξη. Τεράστιε ευκαιρίε και δυναμικό. Να γίνουμε πρωταγωνιστές σε βιομηχανίες με χαμηλή χρήση άνθρακα, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα και ο υπόλοιπος κόσμος θα μας ακολουθήσει. Δεν θα πρέπει να ε, ζητούμε μόνο οι υψηλότερε δεσμεύσει στο Παρίσι, αλλά να αναπτύξουμε και νέες τεχνολογίες. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη που σας κόβω, αλλά είναι οι δημοκρατικοί κανόνες. Αυτοί να τηρούμε το χρόνο. Η κυρία Τερέσα Γκρίφιν είναι η επόμενη. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε. Πουλήσατε βέβαια τις μετοχές σας πρόσφατα, παρόλα αυτά ήσασταν πρόεδρος των εταιριών αυτών και δημιουργήσατε στενές διασυνδέσεις με την πετρελαϊκή βιομηχανία. Πώς θα είσαστε αντικειμενικός λοιπόν στο μέλλον, στο ρόλο σας απέναντι στη βιομηχανία. Δεύτερον, σε πολλά μέρη της Ευρώπης η ενέργεια κοστίζει όλο και παραπάνω κάτι που πιέζει πάρα πολύ τους πιο ευάλωτους και τους πιο φτωχούς της κοινωνίας μας. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να είναι αναγκασμένος να διαλέξει κατά πόσο θα ζεσταθεί ή θα φάει. Τι συγκεκριμένες προτάσεις λοιπόν θα υποβάλλετε ως Επίτροπος για να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό της ενεργειακής ένδυας. Τέλος, μπορείτε να διευκρινίσετε λιγάκι τα σχόλιά σας στο όταν λέτε ότι είναι δύσκολο να συζητήσουν άντρες με γυναίκες επειδή έτσι η πνευματική υπεροχή των ανδρών είναι σε βάρος των γυναικών. Απάντηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητάω με γυναίκες. Είπα εξάλλου στην αρχή ότι ήταν λάθος το σχόλιο μου αυτό και ζήτησα συγγνώμη. Ήτανε σφάλμα. Ζήτησα συγγνώμη, αλλά βλέπετε ότι συζητάμε, το συζητάμε χωρίς πρόβλημα. Τώρα για τις πιο σχετικές ερωτήσεις σας. Ανεξάρτητος ήμουνα πάντα στη ζωή μου. Και όντω ήμουν ιδιοκτήτης αυτών των πιο διάσημων μετοχών της Ευρώπης, έτσι. Αλλά ήμουνα και στο Green Group εκείνη την εποχή ήμουνα υπέρ της πράσινης ενέργειας. Αυτή ήταν η θέση μου. Και ζητούσα φιλόδοξους κλιματικούς στόχους και στήριζα την καθαρή ενέργεια. Το έκανα στο παρελθόν, θα το κάνω και στο μέλλον. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα συμφέροντά μου και αν υπάρξει κάποια στιγμή τέτοιο θέμα υπάρχει ο κώδικας διοντολογίας των επιτρόπων. Βάσει αυτού θα πορευθώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Πολύ σημαντικό. Έγιναν προσπάθειες για ένα κοινό ορισμό, για μια κοινή προσέγγιση. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι μέσα στην ενεργειακή μας πολιτική θα ασχοληθούμε με αυτό ή σε διάφορες πολιτικές, κοινωνικές κλπ. Στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής η καλύτερη προσέγγιση είναι να έχουμε ευθύς μετρητές ώστε να μπορούμε να πετύχουμε και καλύτερη τιμολόγηση, να κοστίζει λιγότερο η θέρμανση και να δίνουμε προτεραιότητα όταν ένα κράτος μέλος στηρίζει νέα κτίρια κτλ. να μπορεί να στηρίξει και το πιο ευάλωτο πληθυσμό ώστε να κοστίζει λιγότερο η ενέργεια, φροντίζοντα δηλαδή για καλύτερη μόνωση των κτηρίων κτλ. Έχουμε πάντως πολλές δυσκολίες και χρειάζεται ακόμα στήριξη πρέπει να το σκεφτούμε ακόμα περισσότερο πώς θα δίνουμε αυτή τη στήριξη. Είναι ζωτική σημασία στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Φρανσουάς Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Απλή γυναίκα είμαι και θεωρώ παρόλα αυτά ότι ο κύριος Γιούνκερ είχε δίκιο να σας αναθέσει αυτό το χαρτοφυλάκιο γιατί ε, είστε απόλυτα εξοικειωμένο ε, με τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Και χαίρομαι για τον αποφασιστικό και κατηγορηματικό σας τόνο που δείχνει επιθυμία να πείσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις προηγούμενες ακροάσει δεν είχαμε πάντα την αίσθηση ότι ο συνομιλητή μα είναι απόλυτα ικανό και επαρκή για τη θέση όπω εσεί. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, σε μια οικονομία χωρί άνθρακα, ε, η διαδικασία δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, στις 8 Ιουλίου του 2014 η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αφιερώσει 300 εκατομμύρια ευρώ μόνο σε ένα θέμα, το θέμα της, δέσμευση δέσμευσης και αποθήκευση άνθρακα. Θα το αναπτύξετε αυτό το πρόγραμμα και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ουδέποτε δεν μιλήσατε για την αποθήκευση ενέργειας. Αυτό είναι, αυτό και είναι σημαντικό θέμα. Έχετε το λόγο κύριε Κανιέτε. Θεωρώ ότι το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρακας ε, για πολύ καιρό θα μείνει παρόν στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα και μεσοπρόθεσμα ε, ο άνθρακας ε, και ο λιγνίτης έχουν σημαντική μαρουσία στο ενεργειακό μείγμα πολλών χωρών και για να επιτρέψουμε στις χώρες αυτές να χρησιμοποιήσουν αυτόχθονες χώρες πηγές ενέργειας, άνθρακα και λιγνίτη δηλαδή, θα πρέπει να αναπτύξουμε προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Βέβαια δεν φτάσαμε ακόμη στη φάση εμπορίας διάθεσης στην αγορά. Αλλά από τα έξι προγράμματα που ενέκρινε η Διεύθυνση Ενέργειας από τα έξι προγράμματα που επέλεξε, τέσσερα ε, έχουν ε, ε, αποτύχει, αλλά δύο έχουν μεγάλες πιθανότητες να φτάσουν στην αγορά. Έχουμε και το πρόγραμμα Νέρσιν 1 με 300 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση για την ανάπτυξή του. Και πολλά κρατημέλη είναι υπέρ αυτού του σχεδίου. Κυρίως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αυτό το NERSIN Υποστηρίζει τέτοια προγράμματα και θα προσφέρουν και τεχνολογία που θα την αξιοποιήσουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εγώ θα υποστηρίξω τέτοια προγράμματα, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων και την εξασφάλιση χρηματοδότησής τους. Γιατί σίγουρα άνθρακας είναι σημαντική πηγή ενέργειας. Τώρα, για την αποθήκευση ενέργειας οι σωρευτές είναι δαπανηροί, δεν είναι και πολύ αποτελεσματικοί, δεν είναι εύκολη η αποθήκευση ενέργειας. Έχουμε βέβαια κάποια προγράμματα που προτάθηκαν για αποθήκευση μέσω συστοιχειών. Θα το δούμε. Ίσως είναι χρήσιμα και για τη θέρμανση. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Αλλά χρειάζεται έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο ώστε να μπορούμε να αξιοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες. Ο Γιολάινεν. Μια πολιτική και μια προσωπική ερώτηση. Επανειλημμένα είπατε ότι ως Επίτροπος θα είστε ουδέτερος σε σχέση με τις πηγές ενέργειας για την υδρογμάτωση, την εξόριξη πετρελαίου, τον άνθρακα. Σωστό είναι αν είστε Επίτροπος Ενέργειας, αλλά η Επίτροπος Περιβάλλοντος δεν είναι λάθος. Εάν θέλουμε να είμαστε παράδειγμα, πρέπει να φύγουμε από τις παλιές ενέργειες, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τις περιορίσουμε. Οπότε έχετε μια πολιτική σύγκρουση συμφερόντων. Και ε, θεωρώ ότι συχνά μπορεί να είστε στη λάθος πλευρά όταν τα λόμπι είναι πολύ ισχυρά. Προσωπική ερώτηση. Προσωπική ερώτηση μετά την πολιτική. Προσωπική. Ε, αναφερθήκατε στον κώδικα δεοντολογίας όπου λέει ότι και προσωπικά και οικογενειακά πρέπει να είστε χωρίς συμφέροντα. Ισχύει ότι ο γαμπρός σας είναι ενεργός στην βιομηχανία πετρελαίου. Και τι θα πείτε στον ε, κύριο Γιούνκερ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, παρακαλώ. Κύριε Λάινεν, όταν ε, μιλούσα για την ε, πυρηνική ενέργεια και την υδρορογμάτωση, είπα για την πυρηνική ενέργεια η υποχρέωσή μου είναι να υπάρχει πυρηνική ασφάλεια, να διασφαλιστεί πυρηνική ασφάλεια με βάση τι υψηλότερε προδιαγραφέ ασφαλεία για του Ευρωπαίου πολίτε. Αυτή είναι η δέσμευσή μου. Για την υδρορογμάτωση είναι αποφάση των κρατών μελών. Η Επιτροπή έκανε συστάσει. Αν χρειαστεί, θα προχωρήσουμε και στην ε, επιβολή κανόνων. Αν χρειαστεί. Τώρα για τη σύγκρουση συμφερόντων. Κοιτάξτε, θα είμαι απόλυτα διαφανή. Θα δείτε και στην ιστοσελίδα μου, εάν γίνω επίτροπο, όλε τι συναντήσει που έχω κάνει με όλα τα άτομα, τι εταιρείε, τα λόμπι, Όλα, όλα θα τα βλέπετε, θα δείτε με ποιον συναντώμε και γιατί. Θα είμαι απόλυτα διαφανής. Και σας είπα ότι έχω ήδη πει. Πούλησα τις μετοχές μου παρά το ότι δεν συνιστούσαν σύγκρουση περιβάλλοντος γιατί σας είπα τι εταιρεία ήταν. Ήταν μια εταιρεία επιμελητίας και αποθήκευσης. Ούτε η ε, γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε εγώ έχουμε την παραμικρή μετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία. Και εγώ θα εργαστώ για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Θα αναπτύξω καθαρέ ενέργειε και για την ε, περίπτωση του άνθρακα. Ανησυχώ, γιατί υπάρχουν χώρε όπω η Πολωνία που έχουν ουσιώδε πρόβλημα. Πρέπει να αναπτυχθεί η δέσμευση και αποθήκευση για να μπορέσουν να διατηρήσουν την παραγωγή ενέργειας μέσω του άνθρακα. Θα στηρίξω λοιπόν τις πιο αποδοτικές τεχνολογίες γιατί το ενεργειακό μείγμα δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Ο άνθρακας θα συνεχίσει να είναι πολύ σημαντικός. Στο μέλλον να περάσουμε σε καθαρότερες ανανεώσιμες. Αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να γίνει αυτό και εντωμεταξύ θα υπάρξει νομοθεσία για να έχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές για την πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Και Τελευταίος, ο Herbert Royal. Παρά την ε, εντύπωση που προσπαθούν να δημιουργήσουν ορισμένοι, δεν είναι εκπρόσωπος των πετρελαϊκών εταιριών, αλλά ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που είχε μια εταιρεία με 50 εργαζόμενους, 50, 5-0. Καμία σύγκρουση συμφερόταν, αλλά παρόλα αυτά σωστά πούλησε και εκείνος και τα παιδιά τους τις ε, μετοχές τους. Δεν ήταν αναγκαίο να το κάνουν. Τώρα μιλάτε για τη γιαγιά του, τον κουνιάδο του. Δεν νομίζω ότι το παρακάνετε. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι είναι δίκαια. Δεύτερον, δεύτερον, δεύτερον. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις παρακαλώ. Κύριε υποψήφια επίτροπε. Πώς, πώς, είπατε ότι μπορείτε πολλά να κάνετε αλλά πώς θα συνδυάσετε την ασφάλεια και τον ανταγωνισμό και την ε, πολιτική για το κλίμα. Τι μπορεί να κάνει ο Επίτροπος για να μην έχουμε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ για το τελευταίο τμήμα της ερώτησής σας. καλοκαίρι έγιναν διάφορες δοκιμές αντοχής μετά την κρίση με την Ουκρανία για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με υπόθεση εργασίας ότι θα σταματούσε η ροή φυσικού αερίου. Και ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δοκιμές για να δείξουν ότι αυτές οι αμφίροπες ροές υπάρχουν, οι αμφίδρομες, ότι έτσι θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Στο μέλλον όμως, Πρέπει να διαφοροποιήσουμε οπωσδήποτε τις πηγές ανεφοδιασμού μας. Με το νότιο διάδρομο, με ανάπτυξη καλύτερων διευκολύσεων hubs, λιμένων, αλλά προκειμένου να είναι ανταγωνιστική βιομηχανία αυτή, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, δίνοντας δωρεάν δικαιώματα, αλλά και με μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί καλά μια εσωτερική αγορά, δηλαδή όπου να υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός και όπου οι τιμές είναι ίδιες ουσιαστικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου θα έχουμε διαφοροποίησει τις πηγές ενέργειας και θα χρησιμοποιούμε περισσότερο τις αναλλακτικές πηγές ενέργειας και θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση της ενέργειας για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια. Είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και όσον αφορά την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Θα αναπτύξουμε επίσης καλύτερες τεχνολογίες για τις αναλλακτικές πηγές ενέργειας και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Η ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή συνδέονται και θα αποτελέσουν μια σημαντική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, υποψήφιε Επίτροπε, για τις απαντήσεις σας. Έληξε λοιπόν το τμήμα ερωταπαντήσεων της ακροασίας μας. Παρακαλώ μια σύντομη παρέμβασή σας, κύριε υποψήφιε Επίτροπε, για να